Συνάδελφοι, παρακαλώ, ας ε, ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Όταν είσαι και εσύ έτοιμος, Μάθιου, θα ήθελα να σας συστήσω, αν και δεν χρειάζεται, τον παλιό μας φίλο και γνώριμο, Τζόρτζ Γιαζεμπόφσκι, που ήρθε να μας ενημερώσει για τα λειτουργικά τμήματα ενέργειου χώρου. Θα θυμάστε ότι είχε έρθει και πέρυσι το Σεπτέμβριο ο Τζόρτζ για μια ενδιάμεση έκθεση, τώρα θα μας ενημερώσει ακόμη πιο διεξοδικά. Είναι ε, πάντα ιδιαίτερη χαρά για μας ε, να σε υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας, George. Και είσαι ευπρόσδεκτος, είτε έρχεσαι με την επίσημη σου ιδιότητα, είτε ανεπίσημα. Ο Σεφ Παρέστης, George, έχεις το λόγο. Well, thank you, Brian. Uh, dear, parliamentarians, dear ladies. Ευχαριστώ, Brian. Χαίρομαι πραγματικά που είμαι εδώ μαζί σας ξανά. Θα απαντήσω και στις ε, ερωτήσεις σας μετά. Έχω μαζί μου και ένα έντυπο το οποίο σας έχει διανεμηθεί για την ε, πρόοδο σχετικά με τα λειτουργικά τμήματα εναρίου χώρου. Καταρχάς θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις και μετά θα μπω σε λεπτομέρεια για τα επιμέρους λειτουργικά τμήματα εναρίου χώρου για να σας δώσω κάποιες ε, λεπτομέρειες. Είμαι στη διάθεσή σας για όλες τις ερωτήσεις που θα θέλετε να κάνετε. Να σας υπενθυμίσω καταρχάς ότι η πρόοδρος όσον αφορά τα λειτουργικά τμήματα εναρίου χώρου ε, ε, ποικίλει από χώρα σε χώρα και σε γενικές γραμμές η πρόοδος είναι εν γέννη αργή. Γιατί είναι αργή? διότι καταρχάς τα κράτη-μέλη σύμφωνα με την νομοθεσία ΣΕΣ 2 ε, είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν τα λειτουργικά του μετανερίου ε, χώρου μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου του 2012, σε 1,5 χρόνο. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη τα ίδια μέσω του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών είπαν ότι θα έπρεπε να επισπευθεί η διαδικασία. Άρα περιμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί η δημιουργία των λειτουργικών θεμάτων αερίου χώρου πριν από τις 4 Δεκεμβρίου του 2012. Και ε, επίσης Υπάρχουν ε, και τα Υπουργεία Εσωτερικών και τα λοιπά που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Χρειαζόμαστε συμφωνία σε, ε, τρίτα, ε, σε τρία επίπεδα για να ολοκληρωθούν και να εφαρμοστούν αυτά τα ΦΑΜ, τα λειτουργικά τμήματα εναερίου χώρου. Και συμφωνία σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο, συμφωνία σε επίπεδο εθνικών αρχών εποπτείας και σε επίπεδο ε, προμηθευτών ε, υπηρεσιών ε, αεροπλοείας, η ANSP, που θα τους λέμε έτσι από εδώ και πέρα, για χάρη συντομίες. Να σας πω ότι η συμφωνία αυτή χρειάζεται και επικύρωση, αλλά η υπογραφή δεν αρκεί και επομένως θα πρέπει να ε, επικυρωθούν γρήγορα οι συμφωνίες αυτές, οι διακρατικές συμφωνίες, έτσι ώστε να ε, είμαστε πιο αποτελεσματικοί στον έλεγχο του, της κυκλοφορία. κυκλοφορίας. Ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια επιτάχυνση των διαδικασιών. Η Ουγγρική Προεδρία θα κάνει ό,τι ε, μπορεί. Ούτως ή άλλως τα ίδια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο αποφάσισαν να εφαρμόσουν την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη είναι πρωταρχικά υπεύθυνα για να καθορίσουν ε, αυτά τα λειτουργικά τμήματα εναρίου χώρου μέσω αμοιβαίων συμφωνιών. Όταν ε, εξετάζουμε την πρόοδο για τη δημιουργία των FAB, σύμφωνα με τα κριτήρια προόδου θα πρέπει να εξετάσουμε τα συγκεκριμένα γεγονότα, τα συγκεκριμένα στοιχεία και όχι τις γενικότητες. Γι' αυτό προσπαθώ και εγώ να δω τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Γι' αυτό η έκθεσή μου είναι λίγες, σελί, λίγες σελίδες, λίγες γραμμές, διότι αναφέρομαι σε συγκεκριμένα στοιχεία, συγκεκριμένα γεγονότα και όχι σε υποσχέσεις. Κάποιες υποσχέσεις ναι, αλλά όχι πολλές υποσχέσεις. Δηλαδή, αν καταγράψει όλε τι υποσχέσει, θα χάσει την πραγματικότητα. Επομένω, όταν, ε, όταν δούμε το έγγραφο, θα ε, δούμε πιο συγκεκριμένα τέσσερα πράγματα. Καταρχάς θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το γεγονό το κατά πόσον υπάρχει καλύτερη, καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στου προμηθευτέ υπηρεσίε αεροπλοεία. Ε, και γιατί αυτό αποτελεί, αν θέλετε, το κλειδί για την βελτίωση της ε, ενέργειας κυκλοφορίας. Δεύτερον είναι να δούμε πόσο η συνεργασία ανάμεσα στους, ε, στον ενέργειο έλεγχο σε πολιτικό και σε, πολιτι... στρατιωτικό επίπεδο είναι, ε, παρουσιάζει μια κάποια ευελιξία. Επίσης θα πρέπει να δούμε τον network manager, τον διευθυντή του δικτύου. το θέμα εξετάζεται ακόμα και ξέρω, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον David McMillan, τον Γενικό Διευθυντή του, του, Eurocontrol και ελπίζω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν και θα επιστρεφθεί και όλη η διαδικασία διορισμού. Επίσης, το τέταρτο πράγμα είναι να δούμε και τις λεπτομέρειες όχι μονάχα τα μεγάλα θέματα. Ας πούμε, η συμφωνία ανάμεσα στους προμηθευτές ε, υπηρεσιών, ε, ανάμεσα στους ε, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όσον αφορά την κατάρτιση, την κινητικότητα. Επίσης, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά το σχεδιασμό και την εφαρμογή για, τους, για, για, για τον εξοπλισμό. Δηλαδή καλό είναι να έχουμε νέες ιδέες και νέα πράγματα όσον αφορά τον, τον αέριο και ε, κυκλοφορία, τον αέριο έλεγχο και αυτά τα πράγματα να μην τα χρησιμοποιεί κανείς ή ένα φαμπ να τα χρησιμοποιεί και ένα άλλο όχι. Άρα επίσης θα πρέπει να εξετάσουμε και τη συνεργασία ανάμεσα στα αεροδρόμια, διότι η, έννοια του ενιαίου εναέριου χώρου, του ενιαίου ουρανού, είναι από το ένα γκέιτ, από τη μία πύλη έως την άλλη. Δηλαδή δεν θέλουμε το αεροπλάνο να κινείται στο, στους διαδρόμους 45 λεπτά για μία πτήση 30 λεπτών. Επομένως και η διάσταση αυτή του αεροδρομίου είναι κάτι ε, πολύ σημαντικό. Ας δούμε τώρα αυτά τα, αυτά τα λειτουργικά τμήματα, αυτά τα τμήματα. Σύμφωνα με την διαδικασία bottom-up από κάτω προς τα πάνω, τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν με ποιον θα συνεργαστούν. Αν δείτε στο χάρτη, στην πρώτη σελίδα, θα δείτε ότι σαν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορείτε να αναρωτηθείτε πόσο δημιουργήθηκαν αυτά τα λειτουργικά τμήματα. Είναι ε, λογική η κατανομή αυτή. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν ποια κράτη-μέλη θα συνεργαστούν. Και αυτή είναι η φάση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Ξεκινώ με το Ηνωμένο Βασίλειο και το, την Ιρλανδία. Αυτό το ΦΑΜΠ ήταν το πρώτο. Και ξεκίνησε πριν από, ε, από το πριν υιοθετηθεί η νομοθεσία CS2. Ε, όπως το βλέπετε και στη σελίδα 2, ξεκίνησε με το MOU, με ένα, με ένα μνημόνιο συμφωνίας ανάμεσα στην Ιρλανδία και στον Ηνωμένο Βασίλειο. Υπογράφηκε το 2008 και τέθηκε σε εφαρμογή πάλι το 2008. Βέβαια, μια και δημιουργήθηκε πριν από το δεύτερο πακέτο, η συνεργασία θα μπορούσε να ενισχυθεί αλλά με τις νέες εξελίξεις, εξελίξεις τις οποίες συνειδητοποίησα και στο Άμστερνταμ την προηγούμενη εβδομάδα, στις 8 Μαρτίου όταν ήμουν εκεί, ξαφνικά τα οι δύο αυτοί προμηθευτές της, του Ηνωμένου Βασιλείου και της ε, ε, Ιρλανδίας συμφώνησαν με τους αντίστοιχους ε, της Σουηδίας και της Δανίας να κάνουν μια μελέτη και αν η μελέτη είναι καλή για το στόχο αυτό θα υπάρξει μία συγχώνευση ανάμεσα στην Βρετανία, Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία και Δανία. Και αυτό είναι πολύ καλή εξέλιξη. Το λέω, το τονίζω και εγώ στο τέλος σελίδας 2. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι NSPs είπαν ότι είναι καλή συνεργασία, αλλά θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη και να έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο FAB, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία. Πολύ καλή προοπτική και εξέλιξη αυτή. Τώρα για τις, ε, θα δείτε τις λεπτομέρειες στο έγγραφο. Μετά παίρνω στο ΦΑΜΠ Δανίας-Σουηδίας που ήταν το δεύτερο στη σειρά που ξεκίνησε. Έγινε μια κρατική συμφωνία του 2009, τέθηκε σε ισχύ το 2010 η συμφωνία αυτή και εδώ υπάρχουν κάποια, ε, κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Οι δύο ANSPs ε των δύο χωρών ε, δημιούργησαν μία εταιρεία, ε, μία ε, Common Holding Company, που ξεκίνησε να αναλαμβάνει τα καθήκοντα των επιμέρους πολιτικών υπηρεσιών, ε, πολιτικών, υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας. Και με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μια ολοκλήρωση ε, μια ενοποίηση όλων των υπηρεσιών που αφορούν ε, την, ε, την κυκλοφορία. Και εδώ θα πρέπει να δείτε και για το ΦΑΜΠ δανια Σουηδία, θα τα αντιμετωπίζουμε από κοινού, ότι συμφώνησαν με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία να προχωρήσουν από κοινού. Και αυτό νομίζω ότι είναι επίση μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Περνάω στο τρίτο φαμπ, σελίδα 6, είναι σε δύσκολη κατάσταση θα έλεγα το φαμπ αυτό. Είναι σαν να κάνετε σαν να μην το είπα. Είναι το βορειοευρωπαϊκό φαμπ. Δείτε τον χάρτη στη σελίδα 1. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι ξεκινάει από την Ισλανδία, Νορβηγία, ε, Δανία, Εστονία, Λετονία, Νορβηγία και έγινε μια δήλωση το, 2000, Σεπτέμβριο του 2010 που δημιούργησε το ΦΑΜΠ αυτό, όμως βρίσκεται σε κίνδυνο το ΦΑΜΠ αυτά για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αυτή η ομάδα των, της Βόρειο, Βόρειας Ευρώπης έκανε μία μελέτη σκοπιμότητας και εκεί ε, εξετάστηκαν διάφορα σενάρια. Ένα μαξιμαλιστικό και ένα ε, μινιμαλιστικό. Ένα δηλαδή πολύ στενή συνεργασία και ένα λιγότερο στενή συνεργασία. Και στι αρχέ σα αυτή τη συνεδρίαση θα πρέπει, ε, διαρωτήθηκαν αν αυτή η μελέτη σκοπιμότητας είναι αρκετά καλή και όρημη για να την υποβάλουν στι κυβερνήσει του. Οι Δανείοι και οι Σουηδοί είπαν όχι δεν είναι καλή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εξού και επέλεξαν την Ιρλανδία και την, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ισλανδία όμως είπε ότι ε, ας περιμένουμε λιγάκι, διαχώρησε τη θέση της η Ισλανδία και οι υπόλοιποι είπαν ε, ωραία θέλουμε να έχουμε μια χαλαρή συνεργασία, μεν, α, τι να κάνουμε τώρα. Επομένως αυτό το φάμπα της Βόρειας Ευρώπης είναι λίγο μπερδεμένο. Ας δούμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Μετά περνάμε στο επόμενο το ΦΑΜΠΕΚ, δηλαδή Κεντρική Ευρώπης, ΦΑΜΠΑ Κεντρικής Ευρώπης, που είναι η τρίτη κρατική συμφωνία, τρεις κρατικές συμφωνίες έχουμε, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία, Σουηδία και αυτή εδώ, Κεντρική Ευρώπης. Αυτή η κρατική συμφωνία ΦΑΜΠΕΚ υπογράφηκε και όλοι περιμένουν να δουν τι θα συμβεί. οι Εθνικές Αρχές Εποπτείας έχουν υπογράψει το Γενάρη μια, αυτή, της, αυτή της χρονιάς μια συμφωνία, αλλά θα θυμόσαστε ότι όταν έπρεπε να υπογραφεί η Συμφωνία ΦΑΜ 2 Δεκεμβρίου, τα κράτη-μέλη ήθελαν να υπογράψουν και μία δήλωση προθέσεων, διότι η κρατική συμφωνία λέει ποιος είναι υπεύθυνος γιατί, όμως δεν διευκρινίζει πώς θα γίνεται, θα αναλαμβάνεται αυτή η ευθύνη. Εξού και θα πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση και να ληφθεί μια απόφαση μέσω μιας ανακοίνωσης, μιας δήλωσης προθέσεων που προβλέπεται ε, να δημοσιευθεί τον Ιούνιο τρέχοντος έτους. Υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι, κάποιες φήμες που λένε ότι τα κράτη-μέλη εγκατέλειψαν την ιδέα να υπάρξει αυτή η δήλωση, η ανακοίνωση προθέσεων. Τέλος πάντων, <clears throat> η κατάσταση είναι ανοιχτή κατά την άποψή μου. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα απλό πρόβλημα, δηλαδή θέμα ε, στάτους αν θέλετε και συμφωνίας ε, ε, ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Στη Γαλλία υπάρχει νέος, γενικός, νέος υφυπουργός μεταφορών και δεν ξέρω... και δεν ξέρω ακόμα ποια είναι η άποψή του. Πάντως το, μοντέλο αυτού του, της holding company νομίζω ότι είναι ένα καλό μοντέλο. Διότι σαν πρώτο βήμα δεν χρειάζεται να ασχοληθείς για το καθεστώς που θα διέπει μια συμφωνία ή κάποια ε, ένωση που, που θα εφαρμόζει και θα λειτουργεί όλα αυτά τα πράγματα εγώ νομίζω ότι το ΦΑΜΠΕΚ, ο ΦΑΜΠΕΚ, το τμήμα αυτό τέλο πάντων τη Κεντρική Ευρώπης, χρειάζεται έναν οδικό χάρτη, δηλαδή να δει πού θα προχωρήσει. Εγώ είμαι Γερμανός και γνωρίζω το συνταγματικό δίκαιο της Γερμανίας αρκετά καλά ε, και νομίζω ότι τέτοιου είδους ε, λύσει θα λειτουργήσουν, λειτουργούν καλά. Όταν ρώτησα για στο Βερολίνο ε, τι γίνεται με, την, με τον νόμο για την επικύρωση, μου είπαν ότι δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Τώρα, το επόμενο είναι, όχι, είναι για, την, ε, για, την, για τις χώρες της Βαλτικής. Είναι λίγο ασύμετρο, αν θέλετε, αυτό το Φάμπ. Έχουμε την Πολωνία και μετά έχουμε τη Λιθουανία από την άλλη πλευρά. Δηλαδή καμία σχέση όσον αφορά το μέγεθος και τον πληθυσμό ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες. Και όσον αφορά την κυκλοφορία, την αέρια επίσης. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται εδώ. Μου είπαν ότι προετοιμάζουν την, ε, μια κρατική συμφωνία που θα υπογραφεί τον Ιούνιο του 2011. Θα είμαι σε δύο εβδομάδες στην Πολωνία και θα σας πω την επόμενη φορά τι ε, θα συμβεί. Μετά έχουμε αυτό γιατί το ΦΑΜΠΑ για την κεντρική Ευρώπη έγινε μια μεγάλη ε, συνάντηση στη Βουδαπέστη την προηγούμενη εβδομάδα και ε, θα υπογράψουν ένα σχέδιο κρατικής συμφωνίας που είχε προγραμματιστεί η υπογραφή της τον Απρίλιο, τώρα λένε μάλλον για τον Μάιο, μάλλον τον Μάιο και όχι τον Απρίλιο. Θα πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εάν δείτε το χάρτη, αυτό το φάμπο της Κεντρικής Ευρώπης, κατά την άποψή μου θα έπρεπε, που είναι Central Europe και όχι Europe Central όπως είναι το διπλανό, το αριστερό, ε, πιστεύουμε ότι επειδή τα αεροπλάνα μας πρέπει να διανύσουν μεγάλη απόσταση, να δείτε στη σελίδα 20, θα δείτε ποιες χώρες έχουν δεσμευθεί να εφαρμόσουν τα ΦΑΜΠ λόγω των συμφωνιών που είχαμε. Ε, πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο αυτό ΦΑΜΠ, επομένως, θα πρέπει να καλύπτει όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Τα κράτη-μέλη όταν υπογράψουν τη Συμφωνία για την Κεντρική Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσουν όχι μόνο πώς θα λειτουργήσουν ε, το δικό τους λειτουργικό τμήμα, αλλά πώς θα ενσωματώσουν και τις υπόλοιπες χώρες. Γιατί κατά την άποψή μου όντως θα πρέπει να ενωθούν. Και μετά πηγαίνουμε στο ΦΑΜΠ για, για τον Δούναβη, Ρουμανία-Βουλγαρία. Εδώ υπήρξαν κάποιες κινήσεις, κάποιες εξελίξεις, υπογράφηκε μία μάλλον προβλέπεται να υπογραφεί κρατική συμφωνία τον Ιούνιο, όχι δεν προβλέπεται, δεν προβλέπεται ακόμα ε, υπογραφή κρατικής ε, συμφωνίας. Άρα ο Δούναμις ακόμα περιμένει, προγραμματίζει και υπάρχει αυτό το memorandum του 2010 και με βάση αυτό θα προχωρήσουν και εκείνοι. Τέλος θα πάω στη Σόφια και θα δω, κάποιες, δω πώς εξελίσσονται τα πράγματα και αν, και αν εξελίσσονται. Επομένως περνάμε τώρα στο επόμενο φαμπ που είναι η νότιο, νότιο-δυτικό φαμπ, Ισπανία-Πορτογαλία. Θα θυμόσαστε ότι υπογράφηκε στην Μαδρίτη μια συμφωνία ανάμεσα στις εποπτικές αρχές. Ε, προχωράνε γρήγορα, ακόμα δεν έχει υπογραφεί η κρατική συμφωνία, τον Ιούνιο προβλέπεται ότι θα γίνει αυτό και υπάρχει, υπάρχει κάποια κίνηση τέλος πάντων. Και επίσης το FAB αυτό θα καλύψει και το Μαρόκο, διότι αν δείτε τον χάρτη θα δείτε ότι υπάρχουν και κάποια νησιά της και της Ισπανίας και της ε, Πορτογαλίας που είναι στα νυχτά του Μαρόκου. Και μετά έχουμε το τελευταίο FAB, το πιο προβληματικό, που είναι το Blue Med, Γαλάζια Μεσόγειος. Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, παρα... Ε, εταίροι, αν θέλετε, είναι η Αλβανία, η Αίγυπτος και η Τινησία και παρατηρητές η Ορδανία και, το και ο Λίβανος. Υπήρξαν κάποιες εξελίξεις οι ANSP και των τεσσάρων χωρών είχαν υπογράψει την προηγούμενη χρονιά μία συμφωνία και εκεί τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά σε υπουργικό επίπεδο υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ε, εγώ έστειλα κάποια επιστολή στους υπουργούς μεταφορών τον Οκτώβριο και περιμένω να γίνει μία συνάντηση ε, που έπρεπε να γίνει στην Ρώμη. Ακόμα περιμένω. Λοιπόν, αυτά με μια γρήγορη ματιά είναι τα όσα συμβαίνουν στα διάφορα FABs. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η πρόοδος ποικίλει και ουσιαστικά αλλά και ε, ε, ε, όσον αφορά το σχεδιασμό εμείς σαν Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά τις εξελίξεις και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στα κράτη-μέλη ότι σύμφωνα με την νομοθεσία SES e έχουν δεσμευθεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος αναφορά την ασφάλεια, τον περιβαλλοντικό κίνδυνο, ε, το κόστος είναι μεγάλες προκλήσεις αυτές και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε αυτό στα κράτη-μέλη και αν τα κράτη-μέλη ε, το ξεχνούν ε, θα πρέπει να τα ταρακουνήσουμε. Και με την περίφημη αυτή εργαλειοθήκη νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε στο τέλος του έτους. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιστροφής που με βοήθησαν και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί είμαι ε, μόνος μου και γι' αυτό η γραμματεία πραγματικά ήταν, ε, με βοήθησε, ήταν πολύτιμη η συνεισφορά της. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Well, thank you very much, George, for that. Ευχαριστούμε πολύ, George. Θα περάσουμε τώρα στο γύρο σχολείων και ερωτήσεων. Έχουμε ένα μισάωρο περίπου για τις ερωταπαντήσεις. Μην το ξεχνάτε. Πρώτος ο κύριος Γκρός. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, vielen Dank für die Präsentation. Also Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γιάννη Μπουζεμπόφσκι για όλες τις ε, πληροφορίες που μας έδωσε. Περιμέναμε πραγματικά από τα κράτη-μέλη να μην κάνουν αρκετά σε αυτού του τομεί και ε, βλέπω ότι πολλοί συνάδελφοι ετοιμάζονται να υποβάλουν σύνδεση ότι που υποβάλαμε ήδη, δηλαδή ποιε είναι οι επιπτώσει των μέτρων μετά τη κρίση που γνωρίσαμε πέρσι στον ενέργειο χώρο. Τελικά βλέπουμε ότι δεν γίνονται αρκετά. Παρόλο που όλες οι χώρες ποια φορά έχουν υπογράψει ότι θέλουν αυτό τον ευρωπαϊκό ένα αεριοχώρο, τον ανοιχτό ουρανό κλπ. Τώρα βλέπουμε ότι δεν γίνονται όσα θα πρέπει να γίνονται. Εάν περιμένουμε μέχρι τα τέλη του έτους, θα έχουμε χάσει νομίζω την προθεσμία του Δεκεμβρίου 2012. Γι' αυτό θα ρωτήσω και την Κομισιόν. Κατά πόσο θα ήταν κατάλληλο το δεύτερο εξάμεινο 2011 αυτό το, αυτά τα εργαλεία, αυτό το toolbox που ανέφερε και ο, ο, Γιώργος να τα ε, εξετάσουμε. Ίσως τελικά καταφέρουμε να αντί να έχουμε μια κόκκινη κάρτα, έχουμε μια κίτρινη κάρτα μόνο. είναι σημαντικά να ξέρω ο συντονιστής πού βλέπει να υπάρχουν τα ουσιαστικά προβλήματα. Είναι θέμα προσωπικού, είναι θέμα τεχνικής συνεργασίας. Και ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες. Και τελευταίο ερώτημα. Αφορά τη σύνθεση των FAB. Ίσως θα βοηθούσε να υπήρχαν ήδη τώρα προτάσεις για διαφορετική σύνθεση γιατί ξέρουμε ότι τα ΦΑΠ δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τα πιο αντικειμενικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια φιλικών σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Ίσως θα μπορούσε από πλευρά συντονιστή και με υποστήριξη του Κοινοβουλίου να υποβληθούν άλλες προτάσεις, χωρίς βέβαια να καθυστερήσει λόγω των προτάσεων το σύνολο της εφαρμογής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο έχει το Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Γιαζεμπόφσκι για την ενημέρωση που μας έκανε, αλλά και για το έργο που έχει μέχρι στιγμής επιτελέσει. Συνεχίζοντας αυτά που είπε ο Ματιέ, διαπιστώνουμε ότι έχουμε μακρύ δρόμο ακόμη μπροστά μας και διαρωτώ με αν μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους είναι δυνατόν να έχουμε κάποια απτά αποτελέσματα. Συμφωνώ με τον Τζόρτζ ότι θα πρέπει να περιμένουμε τα τέλη του έτους για να παρατρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση. Όλοι από κοινού μπορούμε να ενισχύσουμε την πίεση μας και προς τα κράτη-μέλη για να επιταχύνουν το ρυθμό τους. Απότερος σκοπός μας είναι να γίνουμε επιτέλους λειτουργικοί σε αυτά τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου. Και αν τα καταφέρουμε θα έχουμε θετικό αντικτύπο και για την οικονομία και για την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του εναέριου χώρου και ούτω καθεξής. Έχω δύο-τρία σχόλια. Καταρχήν, συμφωνώ με τον κύριο Γιωσεμπόφσκι ότι οι υπογραφές είναι σημαντικές, αλλά το πιο σημαντικό είναι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων το λειτουργικό σκέλος δηλαδή. Πρόσφατα σχετικά, ένα τμήμα των, των κονδυλίων το αφιερώσαμε στην καλύτερη διαχείριση των FAB. Πιστεύετε ότι χρησιμοποιούνται, μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά αυτά τα κονδύλια. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Υπάρχει το θέμα του καταστατικού, έχουμε διαφορετικές ιστορικές παραδόσεις και εκεί έχουμε ένα επίμαχο ζήτημα. Προτείνεται ως μεταβατικό μέσο τη σύσταση ενός holding. Καλή ιδέα αυτή και με τον κύριο Γκρός το είχαμε συζητήσει. Μάλιστα ο κύριος Γκρός αναφέρθηκε και στη Eurocontrol. Και εκεί παρόμοιο πρόβλημα έχουμε με προσωπικό που είναι αποσπασμένο από διάφορες χώρες μέλη. Και πολλές φορές οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, αλλά τελικά καταφέραμε να καταλήξουμε σε καταστατικό που τη χάνει γενικής αποδοχής. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει την πίεση προς τα κράτη-μέλη, με τη δική μας φυσικά βοήθεια. Δεύτερον, Πώ χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια που απελευθερώσαμε. Υπάρχουν ήδη κάποια αυτά αποτελέσματα. Και τρίτο ζήτημα του προσωπικού. Μήπω μπορούμε να εμπνευστούμε από τη Eurocontrol για να επιλύσουμε το θέμα του προσωπικού και εκεί. Κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ. Έχω και κάτι άλλο να σα πω. Για δεύτερη φορά, και σήμερα το πρωί δηλαδή, δεν έχει φτάσει ο καφέ εδώ. Γιατί η δουλειά μα ίσω δεν είναι πάρα πολύ αποφασιστικό. Για μένα προσωπικά όμω είναι. Για να ξυπνήσω. Λοιπόν, αυτό εισαγωγικά. Ξέρω, εσείς έχετε καφέ. Ε, δεν ήρθε κανένα όμω δεν έφτασε μέχρι εμένα κανένα. Ε, μην ανησυχείτε, θα φροντίσουμε. Εγώ προσωπικά θα σας φέρω καφέ. Δεν ήταν βέβαια το πιο σημαντικό, αλλά θεώρησα ότι θα πρέπει να το πω για να μην γίνεται κάθε φορά το ίδιο. Ωραία. Ευχαριστώ τον ε, κ. τον συντονιστή μας για το ΘΑΠ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ελέγξαν ήδη. Περιμένουμε τον ενιαίο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που ελέγξαν για να είναι δυνατή η μεταφορά από τη μια άκρη της Ευρώπης στην άλλη χωρίς προβλήματα. Θεωρητικά γίνεται, στην πράξη όχι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το να υπογραφούν ε, κάποιες συμφωνίες είναι το ένα, η εφαρμογή άλλο. Τι γίνεται, μέχρι τα τέλη του 2012 θέλουμε να έχουμε τελειώσει. Αλλά δεν νομίζω να τα καταφέρουμε, γιατί μόνο οι υπογραφές ακριβώς δεν αρκούν. Και πολλοί διαφανούν, λένε ότι θα πρέπει να ξαναεκπαιδευτούν όλοι οι ελεγκτές ενεργού χώρου για να ξέρουν καλύτερα τις νέες, τους νέους διαδρόμους που είναι πιο αποτελεσματικοί, οι φιλιακοί προς το περιβάλλον, εξοικονομούν καύσιμα κλπ. Πώς θα μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα. Πότε θα μπορούμε να έχουμε επιτέλους αυτόν τον ενίο ευρωπαϊκό χώρο. Στο ΦΑΜΠΕΚ ας πούμε. Με τριοπαθός. Θα ήταν για μένα πολύ ενδιαφέρον. Και κατόπιν ε, πολλοί πολίτες με ρωτάνε θα πρέπει να αλλάξουν όλοι οι διάδρομοι και οι διάδρομοι προσγειώσεως και προσέγγιση του αεροδρομίου κλπ. Όχι. Δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει και θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λίχτινμπεργα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, σε λεπτομέρειες. Από ό,τι θυμάμαι υπήρχε πάντα μία δυσκολία με την ξένηση εκείνη για το Καλίνιγκρατ. Τι γίνεται τώρα. Γιατί υπάρχει ένα πέρα με τον Ρώσο εταίρο μας βέβαια. Και ο, το ΦΑΠ επίσης Κεντρικής Ευρώπης Κάπω περίεργο είναι. Γιατί κοιτάω τι γίνεται στη Μεσόγειο, παραδείγματο χάρη. Ε, συμπεριλαμβάνεται η Κορσική. Και μετά ένα κομμάτι κατεβαίνει προς τα κάτω που δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Ή σχετίζεται με παραδοσιακά μπλοκ ενέργειου χώρου που τα έχουμε αναλάβει δηλαδή από το παρελθόν. Βόρειο ΦΑΠ τώρα. σε ένα με ενό μεγάλου τμήματος του Ατλαντικού ή τη Βορειοθάλασσα. Τα στρατιωτικά συμφέροντα είναι αντίθετα προς την αυτή καλύτερη μορφή νομίζω ή όχι. Και τελειώνοντας. Ένα από τα επιχειρήματα κατά είναι τα προβλήματα προσωπικού στα διάφορα κράτη-μέλη. Τι γίνεται τώρα. Γιατί στην αρχή η Κομισιόν έριξε ένα πετραδάκι στη λίμνη και άρχισε να, κάνει αυτό μεγάλο κύκλο και ελέγχει τώρα ότι θα πρέπει να γίνουν πολλέ εξοικονομίε προσωπικού τι γίνεται ακριβώς. Και το τελευταίο που θυγανίζει με αυτά που ελέγχθησαν ήδη. Παρό λέγεται θα έπρεπε, θα έπρεπε αυτό, θα έπρεπε εκείνο, θα πρέπει να τελειώσει, θα πρέπει να ολοκληρωθεί, θα πρέπει να υπογραφεί. Για την συγκεκριμένη πραγματοποίηση υπάρχει μια δυνατότητα να έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα με το 2012. Τι θα είναι δηλαδή λειτουργικό πραγματικά μέχρι το τέλη του 2012. Ή ποια θα είναι τα μέτρα που θα βελτιώσουν την κατάσταση και κάτι επίση που μου λείπει που υπάρχουν ακόμα οι δυσκολίες με τον στρατιωτικό αέριο χώρο όπως σας είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φώστερ. Um, thank Ευχαριστώ, Γιώργ, γιατί πραγματικά ήταν διεξοδική η παρουσίαση που μας έκανε και ελπίζω να προλάβω κάποια στιγμή να μελετήσω πιο αναλυτικά και το φυλάδιό σου. Ξέρω ότι έχει τριμώξει πολύ κόσμο και το λέω φυσικά μεταφορικά προσπαθώντας να τους παρατρύνεις να σημειώσουν πρόοδο και εγώ υποστηρίζω την ε, προσπάθειά σου. Αναφέρθηκες στην χρήση ενέργειου και ε, πολιτικού και στρατιωτικού ενέργειου χώρου και την ελαστική χρήση που εφαρμόζουν ορισμένε χώρε, το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ άλλων. Κάτι που διευκολύνει και την εφαρμογή των ΦΑΒ, αυτών των λειτουργικών τμήματων ενέργειου χώρου. Γιατί για ορισμένε χώρε υπάρχει πολιτικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τη χρήση του στρατιωτικού ενέργειου χώρου και του πολιτικού. Σε μερικέ χώρε είναι εθνικό το πολιτικό ζήτημα και ελπίζω παρόλα αυτά να σημειωθεί πρόοδο. Σε ό,τι αφορά την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και το ΦΑΠ τους που ανέφερε, φυσικά ω Βρετανίδα χαίρομαι για το πώ έχει προχωρήσει αυτό το θέμα και υπήρχε και στενή συνεργασία και στο παρελθόν πριν την συζήτηση για τα ΦΑΠ Τώρα έχουμε ε, συζητήσεις και με το δανό-σουηδικό ΦΑΠ και μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ε, και μέλος του ΝΑΤΟ και εκεί υπάρχει συνεργασία με τις σκανδιναβικές χώρες. Φυσικά, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει τεράστια προθυμία κάποιων χωρών, αλλά Όλα αυτά τα χρόνια κάναμε τεράστιες προσπάθειες να μειώσουμε και τις εκπομπές, τις καθυστερήσεις και το 90% του ευρωπαϊκού, ε, της ευρωπαϊκής ενέργειας κυκλοφορίας περνάει από το Βόρειο Ατλαντικό και χρειαζόμαστε τέτοιες βελτιώσεις στην Ευρώπη γιατί έχουμε πραγματικά συμφορήσει εκεί, γι' αυτό και χρειαζόμαστε τα FAB κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ήδη ξεκίνησαν κάποιες ε, θετικές πρωτοβουλίες ε, για το περιβάλλον και γίνεται προσπάθεια για να περιορίσουμε και τις εκπομπές ε, του διοξιδίου του άνθρακα και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται. Υπάρχει το θέμα του σχεδιασμού, το διασυνοριακό και το Λονδοχύθρο με τις ε, ε, ε, αναχωρήσεις από το βόρειο, πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι εκεί που σημειώθηκε πρόοδος είναι απτά τα αποτελέσματα και ελπίζω τα κράτη-μέλη, γιατί μερικές φορές είναι περίπλοκη κατάσταση, που διστάζουν να πιστούν. Και τελικά θα ευνοηθούν και οι επιχειρήσει γιατί μειώνεται και το κόστο στη τελική ανάλυση με τα λειτουργικά αυτά τμήματα. Γιώργ, μίλησε για ένα είδο ε, ε, ενοποίηση των προμηθευτών υπηρεσιών αεροπλοεία. Βέβαια δεν, δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση ακόμα μεταξύ των ΝΑΤΣ και της IAA. Δεν είναι προϋπόθεση για τα FAB. Πάντως, καλό είναι που δίνεται έφαση και στο Σέζαρ, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια όθηση προς τα κράτη-μέλη να, να προωθήσουν το Σέζαρ ούτως άλλως. Συγχαρητή, λοιπόν, έχει την αμέριστη υποστήριξή μας και όπως είπα υπάρχουν κάποια παραδείγματα θετικά, ώστε ακόμη και τα κράτη-μέλη που διστάζουν να ενθαρρυνθούν και να αναζητήσουν πιο συγκεκριμένε λύσει. Ευχαριστώ. Κύριος Μαρινέσκου. pentru prezentarea Ευχαριστώ. Έχω ένα σχόλιο, γιατί κοίταξε την έκθεση που μας δώσετε από την προηγούμενη συνεδρίαση και έχω δύο διαφορετικά έγγραφα. Έχω δύο διαφορετικά έγγραφα λοιπόν και προσπαθώ να τα συγκρίνω και βλέπω αρκετές διαφορές. Μεταξύ των δύο παραλλαγών. Έχουν προσθεθεί κάποια ερωτήματα που όμως παρέμειναν αναπάντητα. Nu există răspunsuri Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δίνονται απαντήσει, όπω σα είπα, στι ερωτήσει που προσθέθηκαν. και μάλιστα φαίνεται σε μερικές περιπτώσεις χρειαζόμαστε σίγουρα αποτελεσματικό έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας και διαπιστώνουμε ότι σε ορισμένε περιπτώσεις η μόνη πρόοδος που διαπιστώθηκε ήταν στο σουηδοδανικό FAB που προσπαθούν να έχουν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας. Στα υπόλοιπα ΦΑΠ δεν βλέπω να υπάρχει πρόοδος. Και τώρα διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχουν διαφορετικές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 approach because this is in my opinion the only way to to reach the the single sky wish of especially the European Parliament not of the member states thank you Thank you, Mr. Marinescu, and thank you for... Ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκου και ευχαριστούμε που περάσετε και στα αγγλικά γιατί είχαμε το τεχνικό πρόβλημα και χρειαστήκαμε λίγο χρόνο για να το διορθώσουμε. Και εγώ έχω, George, κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το σχόλιο της κυρίας ε, Φώστερ για την ενοποίηση των ANSP. Δηλαδή, να έχουμε τέσσερα ή πέντε FAB ε, εφαρμόζοντας αυτή την ενοποίηση. Είναι πιθανή μια τέτοια εξέλιξη στο μέλλον και εφικτή. Και όπως είπε και η κυρία Λιχτεμπέργκερ και άλλοι, σε ό,τι αφορά τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας. Υπάρχει μια αντίληψη σε ορισμένες χώρες. These functional airspace blocks will mean job cuts, job losses, Armageddon, uh, the end of the world. How do you think we can try and alleviate those fears uh, and how do you think we can work towards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 starting with, with what, what are the problems? Uh, sorry? Oh, ja, ich spreche Deutsch. Kann ich Deutsch sprechen? Ja, ich spreche Deutsch. Gott. Nein? Was kann ich denn sprechen? So, have we no interpretation at all? Τώρα υπάρχει διερμηνία. Μπορεί να συνεχίσει ο κ. Γρυμπόσκη. Σε ό,τι γλώσσα θέλει. Try again, George, in German. Yeah. Uh, wie sieht das aus, wenn... Άμα μιλάω γερμανικά με καταλαβαίνετε, μεταφράζεται πολύ ωραία. Λοιπόν, θα αρχίσω ξανά για τα γερμανικά, ωραία γλώσσα, που την καταλαβαίνω κιόλα κάπω. Λοιπόν, ερωτήθη ε, κάποιο ε, εάν αγαπάει τη γλώσσα του, είπε εγώ αγαπάω τη γυναίκα μου, τη γλώσσα μου προσπαθώ να τη μιλήσω απλώς. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα εξαιτία των οποίων ε, προχωρούν τα πράγματα τόσο αργά. Πολλά προβλήματα και θα προσπαθήσω να τους σκιαγραφίσω. Σε επίπεδο κρατών υπάρχουν πολλά προβλήματα κυριαρχίας και αρμοδιότητας. Εάν δύο χώρες θέλουν να διπλωματευτούν μεταξύ τους για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ΦΑΜΠ, πρέπει να συνενωθούν οι Υπουργοί Μεταφορών, μετά οι Υπουργοί Άμυνας, μετά οι Υπουργοί Οικονομικών, εάν υπάρχουν κάποια οικονομικά θέματα και σε ορισμένε φορές πρέπει ακόμα και οι Υπουργοί Εξωτερικών να συνεννοηθούν. Τώρα είχα πάει σε μια πρωτεύουσα και μου είπε ο υπεύθυνο για το αεροδρόμιο στο Υπουργείο Άμα θέλω να μιλήσω στη διπλανή αίθουσα με τον συνάδελφό μου, θα πρέπει να περάσω από το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχουν δηλαδή και τυπικά προβλήματα. Και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι λογικό, δεν αρκεί να συμφωνήσει ο Υπουργό Μεταφορών και μετά ο Υπουργό ε, Οικονομικών ή Άμυνα να μπλοκάρει. Θα πρέπει λοιπόν σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου να υπάρχει η συνεννόηση. Και αν έχετε 7-8 χώρες, σε κάθε χώρα τρεις-τέσσερις υπουργοί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι σημαίνει αυτό εν τελευταία αναλύση. Το δεύτερο πρόβλημα. Ορισμένες οργανώσεις ε, ε, ελέγχου του εναερίου χώρου φοβούνται όταν υπάρχουν νέοι διάδρομοι οι νέε νέες περιοχέ θα χάσουν έσοδα. Ποιο θέλει να χάσει έσοδα. Ωραία, να πούμε, θα ελέγχεται διαφορετικά ο χώρο, ο αέριο από χώρα σε χώρα, γιατί αυτό είναι λογικό. Ναι. Αλλά μετά λένε ναι, αλλά 5% των εισόδων μου θα χάσω, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Λοιπόν και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Όσον αφορά το θέμα του καθεστώσεως των οργανώσεων και του προσωπικού. Θα πρέπει νομίζω να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ενδιάμεσα μοντέλα, γιατί δεν έχει νόημα να θέλουμε γλίγορες επιτυχίες και έξι χώρες που έχουν διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης να περιμένουμε να συμφωνήσουν σε ένα μοντέλο. Δεν θα το πετύχουν αυτό σε δύο χρόνια, ούτε καν να συμφωνήσουν και όχι να εφαρμόσουν. Και γι' αυτό είπαμε θα πρέπει να υπάρχει αυτή η εταιρεία, αυτή η holding company, όπου η κάθε οργάνωση ελέγχου του ενωρίου χώρου θα παραμείνει με το δικό της καθεστώς και το δικό της προσωπικό. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πούμε στους ελεκτές ενωρίου χώρου, ότι ακόμα και αν υπάρχει αυτό το holding, θα πούμε, εσύ έχεις όμως το δικαίωμα να παραμείνεις στο δικό σου καθεστώς όσον αφορά τον χρόνο εργά, οργάνωση, το μισθό, τη σύνταξη κλπ. Μόνο άμα τα πούμε αυτά έτσι στους λεκτές αερίου χώρου μπορούμε να τους αφαιρέσουμε το φόβο. Μίλησα την περασμένη εβδομάδα. τους πούμε, δεν χρειάζεται να φοβάσαι να χάσει τη ζωή σου. Για δύο λόγους. Καταρχήν υπάρχουν ελλείμματα ελεγκτών αερίου χώρου. Στη Γερμανία, παραδείγματο χάρη, και δεν είναι η μόνη χώρα. Και δεύτερον, περιμένουμε ότι θα υπάρχει αύξηση των αερομεταφορών και θα χρειαστούν ακόμα περισσότεροι ελεκτέ εναερίου χώρου. Ακόμα δηλαδή και αν εργαζόμασταν πιο αποτελεσματικά που θα το πρότεινα, δεν θα χάσει τη δουλειά του ούτε ένα ελεγκτή. Τον αντίο το είπα στη διάσκεψη στη Βουδαπέστη, θα πρέπει να οργανωθούμε ούτω ώστε να έχουμε μια κινητικότητα για του ελεκτέ αυτού εναερίου Δηλαδή ένας ελεκτής που έχει εκπαιδευτεί σε μία χώρα έχει βέβαια αυτό το πρόβλημα το γνωστό με τη γλώσσα. Το ξέρουμε και από τους αεροδρόμους. Αλλά κατά βάση αυτό είναι δευτερεύον πρόβλημα. Γιατί και το λογισμικό και οι υπολογιστές και το υλικό είναι τα ίδια παντού. Δηλαδή αν είναι κανένας ε, Ελεκτή αερίου χώρου μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ΠΕΤΟΥ Και μια που στον έλεγχο αερίου χώρου η γλώσσα επικοινωνίας είναι πάντα τα αγγλικά, Καλά, θα μπορούμε να πούμε όταν είναι κατα... κάποια καταστροφή μπορεί να τηλεφωνήσει κανείς στην τόπια αστυνομία για να βοηθήσει. Αλλά ακόμα και στη Γερμανία καταφέραμε να μπορούν να εργάζονται τώρα οι Ιταλοί ελεκτές ενεργού χώρου στη Γερμανία χωρίς να κάνουν πέντε χρόνια μαθήματα γερμανικών. Γιατί η κύρια του δουλειά γίνεται με ένα μηχάνημα, με ένα λογισμικό συγκεκριμένο. Αυτό είναι δυνατό νομίζω και το είπα εγώ προς τους ελεκτές. Θα πρέπει να έχετε ίδιο συμφέρον για κινητικότητα. Δεν θέλουν να εργάζονται όλοι στη Βορρή Γερμανία που βρέχει συνεχώ και θέλουν να πάνε στην Ισπανία ας πούμε. Υπάρχουν λοιπόν επιχειρήματα και προσωπικά έχουν κάθε συμφέρον. Εάν λοιπόν συζητήσει κανένα με του ελεκτέ, μπορώ να του το πω αυτό τα πράγματα ξεκάθαρα. Και αν υπάρχει αυτή η εταιρεία holding, μπορεί να κάνει κανεί αυτό για το οποίο υπάρχουν ήδη παραδείγματα. Να πει δηλαδή ότι το υπάρχον προσωπικό παραμένει στο καθεστώς του εκάστοτε. Και ένας κρατικός υπάλληλο εργάζεται δίπλα σε έναν ε, απλό υπάλληλο και δίπλα σε έναν αξιωματικό. Ο καθένας έχει το δικό του καθεστώς, το δική τη σύνταξη δεν χάσει τίποτα. Μπορούν κάλλιστα να συνεργαστούν. Επί της δεν υπάρχουν διαφορές. Είναι θέμα νοοτροπίας, κατά πόσο προτίθεται να το κάνουν αυτό. Σε ορισμένες χώρες η πρόθεση υπάρχει, σε άλλες χώρες δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα που διαβλέπω αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τα FAB, για κοιτάξτε, το πίνακα θα μπορούσα κάλλιστα να φανταστώ. Έχουμε ένα βόρειο τομέα, ένα δυτικό, ένα κεντρικό, ένα κέντρο ανατολικό, κέντρο δυτικό. Βαλτική, Φαψέ και Δόμναβη, ας πούμε, μαζί. Δεν θα ήταν άσχημο. μπορούσαμε από τους 9 να μειώσουμε στους 4-5 και να μειώνουμε όσο πάει περισσότερο τον ρυθμό. Θα πρέπει όμως αυτό το θέμα να μην το υπερβάλλουμε. Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα, το αποφασίζουν αυτό. Μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2012, με διμερείς τουλάχιστον συμφωνίες, είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν ποιος θα κάνει τι με ποιον. Δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε, να τους συστήσουμε, να δώσουμε κάποιες ιδέες, αλλά τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα Και όσον αφορά τις επιστολές αυτές προειδοποίησης, εγώ προσωπικά είπα στον Επίτροπο να αρχίσει να γράφει τι επιστολές αυτές το φθινόπωρο, χειμώνα, κάπου εκεί. Γιατί εάν δεν έχει υπογραφεί καν η κρατική συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτους και επικαιρωθεί, δεν θα πετύχουμε τίποτα μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου του 2012. Αλλά ο Επίτροπος πρέπει να σεβαστεί την νομοθεσία, γι' αυτό τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα καταρχήν, αλλά σας ενθαρρύνω εσείς να μιλήσετε με τις εκάστοτε κυβερνήσεις και να τους πείτε με πού έχετε φτάσει μέχρι στιγμής, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Η συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής αεροπορία έχει δύο πτυχέ. Σε ορισμένε χώρες ο έλεγχος του ενεργού χώρου γίνεται ενιαία. Σε άλλε χώρες υπάρχουν δύο ανεξάρτητες οργανώσεις. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα αν θέλετε να έχουν μια ανεξάρτητη οργάνωση για το στρατιωτικό σκέλος, γιατί αυτή η νομοθεσία εδώ αφορά την πολιτική αεροπορία. Αλλά όπως σας είπα, νομίζω σε ορισμένες χώρες υπάρχει η βούληση με καλύτερη συνεργασία να μελετηθεί το θέμα τους, ε, του κοινού, από κοινού ελέγχου. Το πρόβλημα δεν είναι ο κοινό ή μη κοινό έλεγχο. Το πρόβλημα είναι οι εναέριοι χώροι που αποκλείονται για τις ε, μεταφορές. Παραδοσιακά γίνεται αυτό για ασκήσεις στρατηγικής αεροπορίας. Παραδείγματο χάρη στα γερμανικά, σύνορα αυτό είναι ιστορικής προέλευσης. Κατά πόσο θα πρέπει να παραμείνουν έτσι οι χώροι αυτοί ή θα μπορούσαν να μεταφερθούν. Το σκεφτούμε το θέμα. Μπορούμε να σκεφτούμε κατά πόσον μπορούν οι Σερβικοί να συμφωνήσουν δύο-τρεις χώρους ασκήσεων να τους συνενώσουν. Εμένα μου είπαν κάποιοι αξιωματικοί, ανοιχτά, ότι το πρόβλημα που έχουν είναι ότι δεν πρέπει να τους στείλουμε όλους ε, στη Βόρεια Νορβηγία ή στον Καναδά. Γιατί λέει ότι ε, χρειάζεται να, να πάω γρήγορα, να μπορώ να πάρω από το αεροδρόμιο γρήγορα στον χώρο ασκήσεων. Αν με στείλετε μέχρι τον Καναδά θα έχω αρκετό, αρκετά καύσιμα για να πάω και να έρθω και να κάνω δύο ασκήσεις μόνο. Δεν γίνεται αυτό. Όσον αφορά τους διαδρόμους πτήσεως, σήμερα το πρωί ακριβώς συζητούσαμε με κάποιον που καταλαβαίνει το θέμα. Μπορούμε να έχουμε βελτίωση του δυναμικού με τροποποιημένους ε, διαδρόμους ε, πτήσεως, αλλά η βελτίωση δεν θα είναι πάνω από 5%. Είναι πολύ καλά οργανωμένα τα πράγματα. Τώρα, η διάδρομη προσέγγιση των αεροδρομίων δεν το κάνουμε Θα πρέπει ο καθένα να κοιτάξει τι θα κάνει. Όχι επειδή εγώ είμαι δηλό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το οικονομικό ζήτημα. Γιατί λέγεται συχνά ότι δεν μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η συνεργασία για να υπάρχουν χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό σε μεγάλο ποσοστό είναι δικαιολογία προφάσιν αμαρτίας. Ε, βέβαια, ε, το θέμα είναι ότι με, μια κρατική εγγύηση μπορούν οι διάφορες οργανώσεις να αγοράσουν το λογισμικό που χρειάζονται ή να χρηματοδοτηθούν για μέσω των ε, τελών που πληρώνουν οι αεροπορικές εταιρείες είναι αυτός ένας μηχανισμός που αφορά τα NSP, ότι δεν χρειάζονται συμπληρωματικά χρήματα, ίσως κάποια εγγύηση τραπεζική ή κρατικά χρήματα για νέα κτίρια. Και παραδέχομαι ότι χώρες που δεν είναι ακόμα αρκετά ανεπτυγμένες υπάρχουν χρήματα από τα προγράμματα TNT ε, κλπ. Δεν νομίζω λοιπόν είναι κεντρικό το θέμα των χρημάτων. Τώρα πάλι για το χάρτη αυτό είναι κάπως ανακριβής, αλλά αρκετά ξεκάθαρος. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή ο χώρος, ο αέριος πάνω από τη ανοιχτή θάλασσα ε, διακανονίζεται από το ΙΚΑΟ και γι' αυτό άμα δείτε ας πούμε στο αγγλικό υπάρχουν αυτές, αυτές οι, οι εγκοπές αν θέλετε έχουμε ένα πρόβλημα με τους Ισλανδούς που κάτι προσπαθούν να κάνουν αυτό αλλά εντάξει για τον ΕΦΑΠ εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ένα στρατιωτικό συμφέρον που να παρεμποδίσει η Νορβηγή έχουν αρκετά ψάρια, αρκετά πετρέλαια και δεν ξέρω κατά πόσο θέλω να συνεργαστούν μαζί μας ή όχι. Με καταλάβατε φαντάζομαι. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Καλή είναι Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε έχουμε αρκετά προβλήματα με τη Ρωσία. Εγώ δεν θέλω να πω με το τίποτα για τα δικαιώματα υπέρπτυσης της Ιβηρίας. Τα είπαμε στο παρελθόν όταν προσεχώς πάω στην Πολωνία θα πρέπει να το συστήσω με την κυβέρνηση εκεί ποια είναι η δική τη άποψη. Υπάρχει ένα σχέδιο που διάβασα το Σαββατοκυριακό. Είχε θυμώσει η γυναίκα μου γιατί το Σαββατοκυριακό θα ήμουν και διάβασα 118 σελίδε έρευνα. Ε, ε, Από την Eurocontrol που αναφέρει όλα τα προγράμματα που υπάρχουν ε, Δεν σα το είπα αυτό αναλυτικά, δεν χρειάζεται να σα δώσω τόσε δικαιολογίε κυρία Λίχτενμπέργκερ. μου επιτέθηκε κάποια χώρα και μου είπε ότι δεν καταγράφω τα σχέδιά τη. Και τη είπα εγώ, εντάξει, του απάντησα εγώ, δεν καταγράφω σχέδια. Άμα κάνετε κάτι πραγματικά, πέστε μου το, θα το γράψω. Τα πιο σημαντικά τα έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή του. Όλα τα άλλα τα έχω αφήσει κατά μέρο. Δούναβης. Προσεχώς θα πάω στην ε, Σόφια και θα πάω και στο Βουκουρέστι για να δω τι θα μπορούμε να κάνουμε εκεί. Για την Ισπανία και την Πορτοκαλία το θέμα είναι το Μαρόκο. Στην Blue Med είναι πότε θα καθησυχάσει η Τουνησία, η Αίγυπτος και η περιοχή. Για τον Δούναβη ίσως υπάρχει επιθυμία συνεργασία από την Τουρκία. Πολλά είναι ανοιχτά λοιπόν εδώ. Καν έχει κανένας κατά νου τη Βαλτική, μπορεί να σκεφτεί και τι γίνεται κάποια στιγμή και την Ουκρανία. Αλλά όλα αυτά είναι αρκετά ανοιχτά. Τα ΦΑΠΣ οργανώνονται από τα κράτη-μέλη, μπορούν να συνεργαστούν με τρίτες χώρες, εμείς και εμείς επίσης το προσπαθούμε, αλλά είναι ελεύθερα. Α, και για το Ευρωκοντρόλ. Το Ευρωκοντρόλ από μια διεθνή οργάνωση πέρασε σε μια ε, οργάνωση πρόσφερας υπηρεσιών. Και μπορώ να πω και το λέω και στους Γάλλους εταίρους μου, ότι κάθε φορά που βλέπω ε, κάποιες δομές ε, κρατικού δικαίου, χρειάζομαι κρατικές συμφωνίες κλπ. και Γι' αυτό η ευρωκοντρόλα δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο μοντέλο. Το μοντέλο ενός holding, όπου θα λέγεται ότι οι μέτοχοι είναι όχι οι ιδιώτες, τα κράτη-μέλη. Αλλά η μορφή της οργάνωσης συνεργασία όπως συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων είναι πιο κομψή και πιο εύκολη. Προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Πώς έχει προχωρήσει το θέμα με το ε, υλικό πρόθεση, ίσως θα μπορεί να το εξηγήσει αυτό η Κομισιόν, πρώτα να σας πω τίποτα ελθασμένο και το θέμα του κατά πόσο θα γραφούν επιστολέ ή όχι, το συζητήστε με τον Επίτροπο όταν έρχεται εδώ, γιατί θα πρέπει να το σκεφτεί από μόνο του. Εγώ προσωπικά συστήνω να περιμένετε λίγο ακόμα. Αλλά σας παρακαλώ, μην αφήσετε το θέμα να ξεχαστεί και εγώ δεν θα το αφήσω. Συζητήστε με κάποιες κυβερνήσει που ξέρετε καλά, γιατί νομίζω ότι το σχέδιο αυτό όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια είναι σημαντικό για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, George. Σε ευχαριστούμε, George. Και άλλοι βέβαια ήθελαν να, να λάβουν το λόγο, αλλά έχουμε ξεπεράσει κατά ένα δεκάλεπτο το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε όμως κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει. Σε ό,τι αφορά τα FAP και τα guidance materials, αν θα μπορούσε να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να απαντήσουμε φυσικά. Περιμέναμε απλώς να επιστρέψει στην αίθουσα ο αρμόδιος, ο κύριος Μπάλτουιν. Mr. Chairman, Κύριε Πρόεδρε, σε κατάλληλη στιγμή δυστυχώ έφυγα από την αίθουσα, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το guidance material. Αυτό βγήκε μετά το Δεκέμβριο του 2010 από την έγκριση από την Επιτροπή Εθερών, Θα γίνει νέα αξιολόγηση μετά την ε, θέση ισχύ του εφαρμοστικού κανονισμού, που ελπίζουμε ότι θα εθετηθεί γύρω στον Ιούνιο του 2011. Θα ήταν χρήσιμο συμπλήρωμα σε αυτή τις πίεσεις που θέλει να εφαρμόσουμε ο κύριος Γερσεμπός και στα κράτη-μέλη. Είμαστε ευγνώμονε ε, προς τον κύριο Γερσεμπόφσκι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όλα τα προβλήματα που είχαμε με τα ΦΑΠ θα ήταν ε, τρει χειρότερα αν δεν ήταν τόσο δραστηριο ο κύριος Γερζεμπόφσκι και δεν έκανε τέτοια προσπάθεια. Είμαστε ευγνώμονε, όπω σα είπα και ευχαριστούμε θερμά που οργανώσετε και τη σημερινή συζήτηση. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε George και σε περιμένουμε με δημονία στην επόμενη μα συνεδρίαση. Ελπίζουμε να μην είναι πολύ αργά, να μην περάσει πολύ καιρό. Εν πάση περιπτώσει, είσαι ευπρόσδεκτο όχι μόνο για τι επίσημε επισκέψει, αλλά και ανεπίσημα. Όλοι έχετε το τηλέφωνό μου. Έχετε το, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ό,τι χρειαστείτε με στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ για την υποστήριξη και σας χαιρετώ. Rather belatedly my Κάπως καθυστερημένα και ζητώ συγγνώμη για αυτό από τον κύριο Δεγκράντες Πασκουάλ. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο, την έκθεση δηλαδή του κυρίου Πασκουάλ. Και παρακαλώ το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει την πολύ κακή συνήθεια να ξεκινάει ιδιωτικές συνομιλίες κατά το τέλος ε, της ε, συζήτηση του κάθε σημείου. Το είπα και το πρωί. Λοιπόν, κύριε Τεγκράντε Πασκουάλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να κάνω έκκληση προς, προς την υπομονή σας γιατί Αρχικά το, η έκθεση αυτή αφορούσε τους ερωτές, τώρα ασχολείται με πολύ ευρύτερα ζητήματα. Καταρχήν ξεκινάω την παρουσίαση με την πεποίθηση ότι οι προτάσεις μου είναι κατάλληλες για την υλοποίηση του στόχου που θέλουμε όλοι να υλοποιήσουμε, να βελτιώσουμε δηλαδή στο μέτρο του δυνατού την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία στα πλαίσια της καταπολέμησης και της τρομοκρατίας. Πριν καταθέσω την έκθεσή μου και πριν καταρτήσω το σχέδιο, είχα επαφέ άμεση ή έμεσε με όλου του ενδιαφερόμενου. Καταρχήν, σε πολιτικό επίπεδο, άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του πολιτικού ηθήνοντε, του εμπειρογνώμονε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω ήταν αναμενόμενο, είχα συναντήσει με του κοιόδη ηγητέ και σε κοινέ συνεδριάσει και διμερώ με τον καθένα από αυτού. Έλαβα υπόψη τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή ΕΒΗ και τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, στην οποία μάλιστα είμαι ταυτόχρονα και σκιώδη ηγητή εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Επισκέφθηκα αεροδρόμια και σύγκρινα τις διάφορες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πειραματικό τρόπο. Επιπλέον άκουσα και οργανώσεις του κλάδου για να καταλήξω συμπεράσματα για το ποιες είναι οι ανησυχίες τους και να σταθμίσω τα εύλογα και άνομα συμφέροντά τους. Επίσης είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση και σύσταση. Θα πρότεινα λοιπόν να διαβάσουμε την ε, ε, την έκθεση αυτή, γιατί η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μετά την ε, τρομοκρατική επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα ε, εμπορικό αεροσκάφος και μετά με την ανείχνευση πολλών πακέτων βόμβας από την Ελλάδα ε, χρειάστηκε να γίνουν ε, περαιτέρω προτάσεις και έμεινε παροχημένη η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν στην έκθεσή μου να υιοθετήσω μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Ταυτόχρονα η έκθεσή μου ασχολήθηκε με τα θέματα των σαρωτών σώματος, την ανάλυση των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί για Gel και Spray και τα μέτρα ασφάλειας ό,τι αφορά το φορτίο και το ταχυδρομείο. Γιατί χρειαζόμαστε την έκθεση αυτή. Καταρχήν, ε, η έκθεση δικαιολογείται από το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αμελήσει το θέμα τη ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Και η καταπολέμηση τη τρομοκρατία ήταν και θα είναι πρωταρχικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω φάνηκε και από τη νέα στρατηγική εσωτερική ασφάλεια Ευρωπαϊκή Ένωση και την αναθεώρηση τη αντιτρομοκρατική πολιτική που γίνεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και η έκθεση αυτή προσπαθεί να βελτιώσει την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Από το 2002 και με συγκεκριμένες ε, και απτές προσεγγίσεις υιοθετήσαμε ένα σύστημα ε, αεροπορικής ασφάλειας, ασφάλειας με βάση το οποίο τα κράτη-μέλη χώρισαν αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία. Και μάλιστα ο κανονισμός 300 του 2008 περιγράφει τις διάφορες πτυχές στις οποίες εντάσσονται τα σημεία τη έκθεση πρωτοβουλία, που ασχολείται με τα ακόλουθα σημεία. Πρώτο θέμα, του εισαρωτέ σώματο. Ποιο είναι το ιστορικό. Όπως φαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, η έκθεση αυτή ακολουθεί ένα καθορισμό της Επιτροπής του 2008 που απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θεώρησε ότι δεν πληρούνταν διάφορες προϋποθέσεις όπως ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οι συνέπειες για την υγεία ή η προστασία των δεδομένων των επιβατών. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διασκεδάσει τι αφιβολίε του Κοινοβουλίου, πραγματοποιώντα έναν έλεγχο επιπτώσεων. Σε ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η νέα γενναία των ασαρωτών πληρεί κατά τη γνώμη μου όλε τι προποθέσει. Το θέμα τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, του σεβασμού τη ιδιωτική ζωή, η μη διακριτική μεταχείριση, η εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασία τη ανθρώπινη υγεία, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό και εκτέλεση των πολιτικών τη Ένωση. Όλα αυτά κατοχυρώνονται στο, στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν είναι αρκετά επιχειρήματα ώστε να καταρρύψουμε τη χρήση των σαρωτών αυτών, γιατί οι σαρωτές πληρούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Και τα σύγχρονα συστήματα δεν είναι αυτά που βλέπουμε σε εφημερίδες ή τα περιοδικά από του επικριτέ των σαρωτών. Τα συστήματα που προτείνουν εδώ δεν δείχνουν το ανθρώπινο σώμα, αλλά ένα ανδρίκελο, μια φωτογραφία του επιβάτη με τα ρούχα ή δίνει ένα πράσινο ok όταν ε, ο επιβάτης περνά χωρίς να, να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός. Ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. Είναι ένα θέμα που τη χάνει συνεχούς αναθεώρησης. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια συνολική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Νευρίου του 2010 ε, προστατεύεται για τη νέα τεχνολογία των σαρωτών και μάλιστα θα καταστρέφονται αυτόματα τα δεδομένα μετά την συγκέντρωσή τους για τους στόχους που έχουν προβλεφθεί. Στην περίπτωση των εικόνων, η ανάγνωσή τους γίνεται από έναν, ειδικό, από έναν συγκεκριμένο υπάλληλο του ίδιου φίλου με τον επιβάτη και δεν θα μπορέσει να τις δει κανένας άλλος, δεν θα μπορέσουν να αποθηκευτούν αυτές οι εικόνες και θα καταστραφούν από τη στιγμή που πέρασε ο επιβάτης από το Σαρωτή ή από τη στιγμή που έφυγε από τη ζώνη ασφάλεια και δεν έχει χαρακτηριστεί ύποπτο. Σε ό,τι αφορά τα αεροδρόμια, τα κράτη-μέλη θα καθορίσουν την τεχνολογία που θα επιλέξουν, υπό την προϋπόθεση όμως ότι πληρούνται οι, θε... οι προϋποθέσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την προστασία της υγείας, το ίδιο ισχύει και εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή τη έδωσε στοιχεία για τι διάφορε τεχνολογίε που χρησιμοποιούν τα σκάνερ και μάλιστα αποκλείονται ως, ε, όσα σκάνερ χρησιμοποιούν ακτίνε ισχύ στην απεικόνηση γιατί δεν πληρούν ε, τα όρια τη οδηγία Ευρατόμ και τις, και τις τιμές που αναφέρονται εκεί. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται μόνο από την αστυνομία σε περίπτωση βάσιμη υπόνοιας. Χώρες όπως η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία ή Τσεχία είναι ακόμη πιο φιλόδοξες στην ε, νομοθεσία τους και δεν επιτρέπουν έκθεση των ατόμων για μη σκοπού σκοπούς σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. Και μάλιστα σε περίπτωση που ένας, ένα κράτος ή ένα αεροδρόμιο χρησιμοποιήσουν σαρωτές οπισθοσκέδασης με ακτινεσχή, ε, θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Διάταξη και να δικαιολογούνται από τους να δικαιολογούνται για τη χρήση αυτή από τις δραστηριότητες και ε, τις οποίες χρησιμοποιούνται. Σε ό,τι αφορά τα σκάνερ, είναι πολύ καλύτερα από αυτά που απλώς ανοιχνεύουν μέταλλα. Επιφέρουν ένα, μια προστιθέμενη αξία που οι, οι, οι συμβατικοί σαρωτές ε, δεν την έχουν. Άλλωστε, είναι μέτρα ανάλογα με τον κίνδυνο που προσπαθούν να αποφύγουν. Και μάλιστα θα είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική για τι χώρε. Οι χώρε όμω που εφαρμόζουν ε, και χρησιμοποιούν αυτέ τι τεχνολογίε, θα πρέπει να εφαρμόσουν κάποια ελάχιστα για όρους όρια. Δεν θα είναι υποχρεωτικά αυτά τα σκάνερ για του επιβάτες. Όσοι όμω αρνούν να περάσουν από αυτού του ερωτέ, θα πρέπει να υποβληθούν σε διαδικασίε ισοδύναμη αποτελεσματικότητα. Και πέραμε τώρα στα υγρά σπρέι και επικτώματα, τζέλ. Η έκθεση αναφέρεται και στα υγρά. Για το θέμα αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη την συζήτηση για την, για την νομοθεσία που υιοθετήθηκε σε σχέση με τα υγρά σπρέι και Gel. Είχαμε τον κανονισμό 1546 του 2006 μετά το περιστατικό του Detroit που συνδεόταν με την ιδέα μετατροπής αυτή, αυτής της απαγόρευσης από έναν έλεγχο των υγρών, εφόσον φυσικά είχαμε στη διάθεσή μας ε, τη σχετική τεχνολογία. Και το τονίζω αυτό, εφόσον υπάρχει ε, κατάλληλη τεχνολογία. Το Σεπτέμβριο του 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε στο ψήφισμά του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναθεώρηση της απαγόρευσης του, των υγρών και την ανάκληση του κανονισμού του 2006. Ο τότε όμως Επίτροπος ε, Μεταφορών, ο κ. Ζακ Μπαρό, ε, δεν συμφώνησε με το ψήφισμα και δεν το τροποποίησε την απαγόρευση μεταφοράς ε, υγρών, γιατί κατά τη γνώμη μου η τεχνολογία δεν ήταν σε θέση να ε, εξασφαλίσει κατάλληλο έλεγχο. Και μάλιστα με την υιοθέτηση του κανονισμού 272 του 2009 που συμπληρώνει τις βασικές κοινέ διατάξεις για την ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας, τονίστηκε η ανάγκη εφαρμογής μεθόδων που θα ήταν ικανές να ανοιχνεύσουν υγρά εκρηκτικά το αργότερο στις 29 Απριλίου του 2011. 10 μάλλον, διορθώνει ο μιλητή. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2009 η Επιτροπή, ο Επιτρόπος Ταγιάννη και το Κοινοβούλιο, ο πρόεδρο τη Επιτροπής ε, Μεταφορών, ο κύριος Σίμψον, που δόξα τω Θεώ εξακολουθεί να είναι πρόεδρο τη Επιτροπή, ε, έκαναν μια ανταλλαγή απόψεων και καταλήξαμε στη σημερινή κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τότε κάτι που είχε ζητήσει ο πρόεδρο Σίμψον. Καταρχήν να βελτιωθεί η κατάσταση των επιβατών που αγοράζουν στα duty free και να καταργηθεί η ανάγκη της κατάσχεσης. Έγινε δεκτή η μετάβαση από τρεις σε δύο φάσεις και όλα αυτά περιλήθηκαν στον κανονισμό 297 του 2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως αναφέρω στην έκθεσή μου, είναι δύο οι φάσεις που προβλέπονται στον κανονισμό. Η πρώτη, τις 29 η Απριλίου του 2011, το αργότερο, τα υγρά, σπρέι και τζέλ που αγοράζονται σε σε αεροδρόμιο τρίτης χώρας ή σε αεροσκάφο μη κοινοτική αεροπορικής εταιρεία μπορούν να περάσουν στις ε, περιορισμένες ζώνες ασφάλειας ή σε ένα αεροσκάφος υπό όρου όμω. Δεύτερη φάση, 29 Απριλίου 2013 το αργότερο, όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να ελέγχουν τα υγρά, σπρέι και τζέλ. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας έχει εξακριβώσει ότι υπάρχει κατάλληλη τεχνολογία για την ανείχνευση υγρών εκρηκτικών. Ως εκ τούτου η παρούσα έκθεση διατρανώνει κάτι που ήδη προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, προασπίζοντας την ασφάλεια των ε, επιβατών και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους. Αυτό που ζητούμε είναι απλώς ε, να εφαρμοστεί η εντολή του Κοινοβουλίου, ε, η σύσταση του Κοινοβουλίου, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη τεχνολογία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τελικά δύο λόγια για το φορτίο και το ταχυδρομείο. Με τις πρόσφατες τρομοκρατικές ε, επιθέσεις σε επιβατικά αεροσκάφη, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο άμεσης δράσης για να εντοπιστούν τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα. Είμαι υπέρ της πρότασης ε, τα σύστημα, ότι τα συστήματα ελέγχου θα πρέπει να είναι αναλογικά και ισοδύναμα, να ελέγχονται τα εμπορεύματα που μεταφέρονται αεροπορικά, γιατί το 70% των εμπορευμάτων μεταφέρονται σε επιβατικά αεροσκάφη. Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί το κόστος, το βάρος, το φορτίο και να δυσχεράνουμε τη μεταφορά εμπορευμάτων με τις αεροπορικές μεταφορές. Θα πρέπει να συνδυάσουμε την ασφάλεια με την αποτελεσματικότητα των κανόνων, να γίνει μια ανάλυση του κόστους και του ωφέλους που έχουμε με τα μέτρα αυτά. Συμπέρασμα λοιπόν κύριε Πρόεδρε και θα σας απαλλάξω σε λίγο. Όλα αυτά τα σημεία της έκθεσης για την ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας αντιστοιχούν σε προηγούμενη τρομοκρατική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να εξασφαλίσει την προστασία των πολιτών και να αποτρέψει στο μέλλον τρομοκρατικές ενέργειες. Εκεί στηρίζεται η έκθεσή μου για μια συνολική ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας με τις μυστικές υπηρεσίες, το προσωπικό ασφάλειας και με την πρόοδο της τεχνολογίας που θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις πτυχές και να προλαμβάνουν τους ε, τρομοκράτες που θέλουν ε, να χρησιμοποιήσουν ε, οποιοδήποτε μέσο για να προκαλέσουν φόβο και τρόμο. Θέλουμε λοιπόν διεύρυνση της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς, γιατί γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ για να προστατεύσουμε τους συμπολίτε μας. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε την συμφωνία και νομίζω ότι σε ένα τόσο αξιέπαινο στόχο που είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρου τα προσωπικά και να υιοθετήσουμε μια λύση που μπορεί να μην αποφεύγει το σύνολο των κινδύνων αλλά τουλάχιστον θα τους περιορίσει το ελάχιστο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε διάφορους ε, ε, ομιλητές. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος να προσθεθεί σε αυτό το κατάλογο των ομιλητών. Εάν όχι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κύριε Ράνερ, ήδη συμπεριλαμβάνεσαι στον κατάλογο, για να ξέρω και πόσο χρόνο θα έχει ο καθένας. Για τους σκιώδεις, πέντε λεπτά και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Μάλλον τρία λεπτά για τους υπολείπους. για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να ομολογήσω ότι ε, θα είχα πάρα πολλά πράγματα να προσθέσω. Βέβαια, εάν μπαίναμε σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες θα είμαστε εδώ μέχρι αύριο. Αλλά τέλος πάντων, στη συγκεκριμένο θέμα θεωρούμε ότι έχουμε προχωρήσει ήδη αρκετά έχοντας κάνει τα μισά. Πάντως ο εισηγητής ε, οφείλω να ομολογήσω ότι έχει δράσει με ιδιαίτερη σοβαρότητα αν θέλετε και κατάφερε να ενσωματώσει τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών. να σχολιάσω κάποια από αυτά τα οποία είπε ο κύριος ε, Πασκουάλε. Ε, οφείλω να ομολογήσω ότι ε, συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπε. τονίσω ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία θα πρέπει να ισχύει σε όλη την Ευρώπη πρέπει να γίνεται και σεβαστή. Για ένα θέμα θα ήθελα ίσως να συζητήσουμε λίγο είναι να δούμε κατά πόσον αυτά τα μηχανήματα είναι απαραίτητα, αναγκαστικά. Μήπως υπάρχουν και άλλοι μέθοδοι που είναι εξίσου αποτελεσματικές ε, και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σαν αναλλακτική λύση. Επίσης προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα ατομικά δικαιώματα κτλ. Όλα αυτά είναι μια προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη και αυτό το οποίο προτείνεται πιστεύω είναι ένας δρόμος τον οποίο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κριτική η οποία γίνεται για τα μηχανήματα αυτά, διότι δείχνουν κάποια ε, σημεία του σώματος, ε, τα οποία οι περισσότεροι δεν θα επιθυμούσαν ε, ε, να εμφανίζονται. Επίσης, ε, όσον αφορά την διάρκεια διατήρησης των εικόνων αυτών, δεν θα έπρεπε να διατηρηθούν με όσο το δυνατόν λιγότερο χρονικό διάστημα. Η όλη διατύπωση πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να προσεχθεί, διότι είναι λίγο ασαφής και γενική. Επίσης, όσον αφορά τα εμπορεύματα, Άλλο πράγμα είναι αυτό. Δεν μιλάμε για ε, μεταφορά επιβατών. Έχει να κάνει ε, ε, έχει να κάνει τίποτα με το θέμα αυτό και η μεταφορά των ε, εμπορευμάτων. Επίσης, στην χρηματοδότηση, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, θα έπρεπε κάπου στα εκτιμώντας να πούμε ότι το Συμβούλιο έχει μιλήσει για τη χρηματοδότηση των αεροδρομίων. Κάπου θα πρέπει να το αναφέρουμε. Πρέπει να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, πιστεύω, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στην διατύπωση. Κυρίως όσον αφορά ε, τις ενέργειες του Συμβουλίου. Πάντως, ούτως ή άλλως, πιστεύω ότι ε, το κείμενο που έχουμε μπροστά μας αποτελεί μια καλή βάση για να προχωρήσουμε. Συνοψίζω λέγοντας ότι το σχέδιο σε γενικές γραμμές είναι καλό, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να προχωρήσουμε ε, για περαιτέρω, όμως χρειάζονται και κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες λεπτομέρειες. Επίσης να σας πω ότι θα πρέπει να φύγω γιατί έχω και άλλες επιτροπές που, σας, ε, που παρακολουθώ. Ε, υπήρχε μια μικρή απόκληση από τα πέντε λεπτά τα οποία είχαμε πει. 4.35. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σεβαστώ και εγώ αυτή την, ε, αυτή την προθεσμία που μου δώσατε. Μιλάω γρήγορα, άρα ξεκινάω καλά. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε τον ε, κύριο Λουίς Ντεγκράντες Πασκουάλ ε, είναι καλή η έκθεσή του, ε, το συζητήσαμε και σε επίπεδο σκιωδών εισηγητών. Είναι μια δυνατότητα που προσφέρεται στους επιβάτες Όταν προσφέρεται μια καλή τεχνολογία και μια καλύτερη κανολογία, ε, δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι οι σαρωτές είναι ένα εργαλείο μόνο σε αυτή την εργαλειοθήκη που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν ε, είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Θα, προφανώς θα πρέπει να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή, θα πρέπει ε, να σεβόμαστε την υγεία ε, των επιβατών. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που δεν θέλουν να περάσουν τους ερωτές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Στη Γερμανία ακούστηκε το θέμα αυτό για λόγους ιατρικούς παραδείγματος χάρη. Τέλος πάντων, στην Γερμανία θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία για να ισχύσουν όλα αυτά τα πράγματα και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Επίσης, Υπάρχει κάτι στην έκθεση που δεν καταλαβαίνω. Στην παράγραφο 24 όσον αφορά την εικόνα του σώματος. Η χρήση των εικόνων του σώματος. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση των εικόνων του σώματος. Μιλάμε για ένα σκιαγράφημα, όχι για ολόκληρες εικόνες του σώματος. Αυτές, η, η ολόκληρη εικόνα του σώματος δεν πρέπει να ε, χρησιμοποιείται, δεν πρέπει να υπάρχει καν. Κάτι άλλο το οποίο δεν καταλαβαίνω είναι η απαγόρευση των, της διακριτικής μετα, μεταχείρισης. Μετά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το έχουμε συζητήσει αυτό. Αν θέλουμε να χρησιμοποιηθεί ε, μια τέτοιου είδους τεχνολογία, το πρόβλημα είναι ποιος θα την πληρώσει. Δεν είναι σαφές ποιος αναλαμβάνει το κόστος εάν είναι προ όφελο των κρατών μελών, θα πρέπει να το αναλάβει το κόστο αυτό το κράτο μέλο. Και δεν είναι μόνο το θέμα των σαρωτών, χρειάζονται και άλλα μέτρα συνοδευτικά, μέτρα προσαρμογή. Δεν θα μπορέσουν κάποια αεροδρόμια να χρησιμοποιήσουν αυτή την τεχνολογία. Επίσης, για την ε, ασφάλεια, μέτρα ασφάλειας για τα φορτία. για τα εμπορεύματα, για τα φορτία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ισχύουσα νομοθεσία. Ή τα πράγματα είναι αρκετά αποτελεσματικά. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Προφανώς, να σκεφτούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Τώρα κάθε όμως πακέτο, κάθε δέμα θα πρέπει να ελεγχθεί. Ίσως θα πρέπει για κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση. Κυρία Λίχτενμπεργκ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο, τον Λουίς Γκράντες Πασκουάλο. Υπάρχουν κάποια πράγματα στην εκθέση που αντικατοπτρίζουν και τις προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε. Θα ήθελα όμως να κάνω κάποιες διευκρινήσεις ή να ζητήσω κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχάς, Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν και ούτως ή άλλως μιλάμε για ευρωπαϊκούς κανόνες που θα εφαρμοστούν. Κατά την άποψή μου, Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα έπρεπε ίσως να εξετάσουμε λιγάκι. Κυρίως, ας πούμε, ξεκινάμε με το σημείο 10. Αυτό το οποίο λέγεται εδώ δεν ε, ισχύει για όλους είναι λίγο στατιστική η δήλωση αυτή. Στο σημείο 9, πριν από το 10, που αφορά την κλιμάκωση της τρομοκρατίας. Λέγεται εδώ ότι η κλιμάκωση της τρομοκρατίας απαιτεί από τις δημόσιες αρχές τη δηλήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης τα οποία ζητούν οι δημοκρατικές κοινωνίες. Είναι μάλλον γενική η διατύπωση αυτή. Ίσως θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι εδώ στο σημείο 9. Επίσης, ε, στο σημείο 14 για τα κράτη-μέλη. Τι εννοείται πιο αυστηρά μέτρα, να εφαρμόσουν πιο αυστηρά μέτρα. Τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν αυτά τα αυστηρότερα μέτρα, δηλαδή θα έχουν περισσότερους αστυνομικούς ελέγχους, περισσότερους αρωτές. Τι σημαίνει πιο αυστηρά μέτρα. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Επίσης, για το σημείο 15, Το πρόβλημα δεν είναι η χρήση των σαρωτών του σώματος που πρέπει να γίνεται με τη θέληση των επιβατών, είναι ότι ενημέρωση έχει πάρει ο επιβάτης. Πρέπει να είναι σαφής η ενημέρωση. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε... Όσον αφορά τους συστηματικούς ελέγχους ασφάλειας, μπορούσα να πούμε κάτι άλλο. Θα μπορούσαμε να πούμε έλεγχοι με ακτίνες έχει γίνονται που και που. Και γι' αυτό θέλω να διαγράψω το συστηματικό. Άλλο συστηματικό και άλλον υπάρχει κάποιος ε, κίνδυνος που έχει καθορίσει η αστυνομία. Λοιπόν, να βγάλουμε αυτό την έκφραση συστηματικά. Γιατί αλλιώς κάθε κράτος μπορεί να κάνει ελέγχους δειγματοληπτικούς με ακτίνες. Εγώ ας πούμε πετάω πολλές φορές και αστρίζεται η επιβάρηση με τις ακτίνες στο σώμα μου. Λοιπόν, να βγούμε τελείως από αυτό το τομέα που είναι θέμα της αστυνομίας Drogen, Brand. Σημείο 20. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφερθούμε στο θέμα της ε, αξιολόγησης των ε, συνεπειών. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται σχετικά με την υγεία για να μπορούμε να διασκεδάξουμε τις επιφυλάξει που υπάρχουν. Μετά, αποθήκευση. αυτή. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τους ε, συναδέλφους. Δεν επιτρέπεται επουδενή. Ούτε με μια ρήτρα που να λέει κάποτε θα χρειάζεται. Ναι, αν πούμε κάποτε θα χρειάζεται, θα γίνεται. Λοιπόν, να μην μαζεύονται τα στοιχεία αυτά. Μια μιατιά και τελείωσε. Γιατί αν πούμε εκεί που χρειάζεται η ασφάλεια των εναερίων μεταφορών είναι μία έκφραση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Γιατί αλλιώ μπορώ να κρατήσω το, την εικόνα ένα εξάμεινο για να δω αν μετά από εξάμεινο αυτό είχε ακόμα τον δημοτοδότη, ε, ή όχι. Σπάντα. Σημείο 30. Κώδικα συμπεριφορά. Που πρόκειται να προετοιμάσουν τα κράτη-μέλη από κοινού. Πόσο δεσμευτικό θα είναι ο κώδικο αυτός. Γιατί αν δεν είναι δεσμευτικό, είναι μια δήλωση προθέσεων πάλι. Κόστος. Αναφέρεται στα μέτρα ασφάλεια όσον αφορά τις ε, εμπορευματικέ μεταβάσει. Όχι, όχι καθόλου. Εγώ κοιτάω το ρολόι, ε. δεν το έχω ξεχάσει. Εγώ... Εγώ κοίταξα το χρόνο γιατί πολύ συχνά εσείς ξεπερνάτε το χρόνο. Και φτάνετε τώρα τα πέντε λεπτά. Speak Σας παρακαλώ. Μα δεν μου επιτρέψετε να τελειώσω την τελευταία μου πρόταση. Και αυτό δεν το κάνετε με κανένα. Ο κύριος Βαντάλα, πέντε λεπτά. Voorzitter, ehm, de rapporteur heeft een goede lijn te pakken. Ε, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που ο εισηγητής αναφέρεται στην ανάλυση του κινδύνου και θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Ένα τμήμα της ανάλυσης του κινδύνου θα πρέπει να προϋποθέτει την ε, ε, αξιολόγηση του προφίλ αυτού. Στο σημείο 13 λέγεται αυτό και στη 15 ε, κατά πόσον κάτι τέτοιο είναι εθελοντικό ή όχι. Δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Καταρχήν για τις ακτίνες εχει Δεν θέλω να υπάρχει καθόλου και το ίδιο ισχύει και για το 8 και για το 18, θα πρέπει να είναι διαφορετική η διατύπωση. Να μην υπάρχουν κανένας τύπου σαρωτές σώματος που να χρησιμοποιούν ακτίνες. Πρέπει να τροποποιηθεί αυτό. Κατόπιν. Η απεικόνιση του σώματος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Αυτό ισχύει για το 24 και για το 23 και για το 25 και για το 27 Αναφέρεται ο εισηγητής σε εικόνες και αγραφήματα. Εγώ δεν θέλω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή η διατύπωση των σημείων αυτών. Και μετά όσον αφορά το σημείο 26. Ο κανόνας θα πρέπει να είναι ότι κάθε ταξιδιώτης που περνάει από τον σαρωτή σώματος, αν πει δεν θέλω, θα πρέπει να μπορεί να ελεχθεί διαφορετικά. Ακόμα και ο διαφορετικός τρόπος διαρκεί περισσότερο. Και μία συγκεκριμένη ερώτηση για τον εισηγητή, για το σημείο 41. Εδώ ζητά η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερους ελεγκτές. Σε ποιους ελεγκτές αναφερόσαστε. Μπορεί να μας το διευκρινίσει ο συγγητής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πέντε λεπτά η κυρία Βάης. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής αναφέρθηκε σε πολλά μέτρα ασφαλείας. Εγώ θέλω να περιορίσω τι παρατηρήσεις μόνο σε σώματος και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον αυτό πραγματικά οδηγεί σε περισσότερη ασφάλεια. Γιατί οι σαρωτές σώματος δεν μπορούν παρά να δουν αυτό που είναι στην επιφάνεια του σώματος και όχι αυτά που είναι μέσα στο σώμα. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ακτίνες. Λοιπόν, όποιος ε, κάνει μια προσπάθεια για να, βα... Ε, βάλει ε, στο αεροπλάνο, θα χρησιμοποιήσει άλλες μεθόδους. Αυτός ο, που προσπάθησε να το βάλει στα ίσορουχά του, από που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, δεν θα είχε ανοιχνευτεί με τους ερωτές αυτούς. Και όπως και η κυρία Ριχτεμπέρη και εμείς θα τελείω ε, το συστηματικό έλεγχο σε όλους τους ταξιδιώτες. Μετά, το τι γίνεται με την εικόνα αυτή. Μέχρι στιγμής δεν καταφέραμε ποτέ 100% να προστατεύσουμε τα προσωπικά ε, δεδομένα. Κάθε σύστημα πληροφορικής έχει τη δυνατότητα να τύχει ε, εσφαλμένης, αν θέλετε, πρόσβασης. Όποιος έχει κακές προθέσεις μπορεί λοιπόν να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά και εάν αποθηκεύονται τα στοιχεία τότε είναι εύκολο να, τα, ε, να έχει πρόσβαση σε αυτά και ε, κάποιος ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα και έτσι δεν προστατεύεται ο ιδιωτικό τομέα ε, των ταξιδιωτών και αυτό μου φαίνεται πραγματικά ενάντια της αξιοπρέπειας γιατί δεν πρόκειται για μια απεικόνιση μονάχα του σώματος, αλλά και για ιατρικά ε, μηχανήματα που ενδεχομένω έχουν οι άνθρωποι στο σώμα τους. Ε, καθετήρες, ε, πάνες, προστασία της υγείας. Εάν οι σαρωτές σώματος χρησιμοποιούν γενικά παντού και πάντα, αυξάνεται πάρα πολύ η επιβάλληση με ακτίνες των ταξιδιωτών. 30-300 GHz είναι η έκθεση των ταξιδιωτών, όπως με τα κινητά και με τα μικροκύματα. Αλλά όπως και για τα κινητά υπάρχουν περιπτώσεις επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία. Και τι γίνεται επίσης με παιδιά, με ε, γυναίκες εγγύως ή με αυτούς που συχνά εκτίθενται στις, ε, στην ακτινοβολία αυτή. Ακόμα και το προσωπικό που στέκεται εκεί μπροστά στις, στο μηχάνημα ή δίπλα στο μηχάνημα μπορεί να υπάρχουν και για το προσωπικό επιπτώσεις αρνητικές στην υγεία. και η πιο ελαφρά μορφή θα ήταν η παθητική έκθεση στις ακτίνες αυτές. Παιδιά επίσης γίνεται πολλές φορές επαναλημ... Ε, επαναλαμβανόμενος έλεγχος γιατί θα πρέπει κανένας να είναι ακίνητος μέσα στους ερωτές αυτούς και τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο να μείνουν ακίνητα όλη την ώρα που γίνεται η σάρωση αυτή. Οπότε η εκθεση τους είναι μεγαλύτερη τελικά. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι 100% ασφαλές, ούτε και αεροπορικές δεν είναι 100%. Καμιά φορά υπάρχουν επιτυχείς ε, τρομοκρατικές ε, ε, ενέργεια τι να πούμε, να πούμε ότι δεν θα πετάξουμε πια καθόλου, αλλά το να υπάρχουν αυτά τα πολύ αμφίβολα μέσα και διαδικασίες επειδή κάτι, κάτι έγινε κάποια φορά δεν νομίζω ότι είναι σωστή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Φώστερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή. συμμετείχα στην σύνταξη της γνωμοδότησης Επιτροπής Περιβάλλοντος και εκεί δώσαμε έμφαση στα θέματα υγείας, όπως ήταν αναμενόμενο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ασχοληθήκαμε και με μια, και θέματα που θίξαμε και εδώ. Το θέμα της, της των σαρωτών πιστοσκέδασης και τι εκτινοβολία χρησιμοποιείται είναι σημαντικό είτε το θέλουν τα κράτη-μέλη είτε όχι, αν ξεπεράσουμε το τεχνολογικό επιχείρημα και ο κόσμος ε, πιστεί ότι ό,τι τεχνολογία και αν χρησιμοποιείται είναι ασφαλής, τότε θα έχουμε σημειώσει ένα βήμα πρόοδου για τους αρωτές σώματος ε, ως συμπληρωματικό θέμα. Σε ό,τι αφορά την ακτινοβολία οπισθοσκέδασης δεν νομίζω ότι μπορεί να σημειώσουμε πρόοδο, γιατί ακόμη και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ασχοληθήκαμε με εξαιρέσει. Και διαρωτηθήκαμε τι τροπή μπορεί να πάρει αυτή η συζήτηση. Είτε θα έχουμε ένα συμπληρωματικό εργαλείο για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, οπότε όλοι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν, είτε μόνο ορισμένα αεροδρόμια αεροδρόμια κράτη-μέρη θα το χρησιμοποιήσουν και είναι προαιρετικό, είτε άλλα, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, θα το επιβάλλουν υποχρεωτικά. Αλλά έτσι θα περιπλέξουμε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όσο συζητούμε τόσο χειρότερα περιπλέκονται τα πράγματα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω. Είπα ότι αν ξεπεράσουμε το ζήτημα της τεχνολογίας ε, και φυσικά ασχοληθούμε με τις πολύ σημαντικές εξαιρέσεις, επανερχόμαστε σε κάτι που έχουμε πει πολλές φορές. Αν τα ξεπεράσουμε όλα αυτά τα τεχνολογικά και τις εξαιρέσεις, σίγουρα πανάκια δεν είναι οποιαδήποτε μέθοδος αλλά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και γι' αυτό χρειαζόμαστε καλύτερη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών, κεντρικό σύστημα κράτη θέσεων, το profiling των επιβατών. Η Επιτροπή Περιβάλλοντο είναι υπέρ των profiling των επιβατών. Γιατί από τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τρομοκρατικέ απειλέ, είναι σημαντικό να συντονιστούμε σε όλα αυτά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια. Ο εισηγητή Δεκράντε ασχολήθηκε με το θέμα τη αποθήκευση ή όχι των εικόνων και για πόσο καιρό αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσουμε αν, προ... αν δεν δώσουμε μια απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα. Θα το έχουμε αυτό συμπληρωματικό εργαλείο και θα είναι υποχρεωτικό για όλα τα κράτη-μέλη ή θα χρησιμοποιούνται μόνο από, από όποιον το επιθυμεί. Και φυσικά μόνο αν έχουμε μια τεχνολογία που θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν όλοι και ο κόσμος θα αισθάνεται ασφαλής και προστατευμένος, αν η πρακτική εφαρμογή είναι ασφαλής, αν η κατάρτιση είναι σωστή. Και φυσικά να έχουμε και ένα one-stop shop ώστε όλα τα κράτη-μέλη να ξέρουν που να απευθύνονται και να μην έχουν πρόβλημα με αυτό. Ευχαριστώ τον εισηγητή και περιμένουμε και τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you, Mrs. Runner. Κυρία Ράνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το θέμα αυτό που ε, παρουσιάζει κάθε ένα πολύ δύσκολο θέμα και καταδεικνύει βέβαια και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και εδώ εγώ έχω κατά νου κυρίως τις συσκευές που ακόμα δεν τις έχουμε και που είναι αμφίβολο εάν θα τις έχουμε κάποτε. Υπάρχει προστασία των στοιχείων, υπάρχει το υλικό που χρησιμοποιείται. Δεν μπορώ παρά να ελπίζω, γιατί εγώ σαν μείνουμε πάντα σε μέση οδό, Ελπίζω ότι η εξέλιξη αυτών των ε, συσκευών και σε αποδεκτό κόστος θα προχωρήσουν πολλά τα πράγματα. Οι δικές μου πληροφορίες πάντως λένε ότι ακόμα χρειάζεται πάρα πολλή εργασία. Και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα ασφαλείας μόνο με στους ε, σώματος. Εάν πολλοί δηλαδή αρνηθούν τον σαρωτή σώματος, θα σταματήσουν θα, θα, θα διακοπεί τελείω ε, η επικοινωνία στο αεροδρόμιο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πιο ευρύς ιδέες ασφάλειας. Δηλαδή το να εξετάσουμε μόνο το θέμα των σωματών σώματος και να μην σκεφτούμε όλα αυτά που υπάρχουν στα περίγυρα, θα οδηγήσει ίσως σε προβλήματα που δεν θα πρέπει να έχουμε και ελπίζω ότι θα ξέρουμε κάτι περισσότερο για τις συσκευές αυτές μέχρι να ολοκληρωθεί το θέμα και τότε να μπορούμε να κάτι να σε Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και Δανέλης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Ντεγκράντες για τη σοβαρή δουλειά που έχει κάνει. Ε, για τα μέτρα ασφάλειας για το φορτίο δεν έχω καμία επιφύλαξη. Είμαι όμως εξαιρετικά ανήσυχος για τα ζητήματα των σαρωτών σώματος, ε, όχι μονάχα για τα θέματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του σεβασμού της αξιοπρέπειας του ατόμου, που ίσως η καινούργια γενιά των σαρωτών έχει κάνει πρόοδο σε σχέση με τους αρχικούς, όμως παραμένουν αναπάντητα αρκετά ερωτήματα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι το ζήτημα παραμένει εντελώς θολό είναι στα θέματα προστασίας της υγείας. Ε, και όσον αφορά τις δύο βασικές τεχνολογίες, δηλαδή το Active Millimeter Wave ε, δεν πάβει να είναι μια καινούργια τεχνολογία οι κίνδυνοι της οποίες για το ανθρώπινο DNA δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς και αυτό μας λένε όλοι οι ειδικοί επιστήμονες. Όσο δε την, ε, για το backscatter X-ray, νομίζω ότι τα πράγματα είναι απολύτως σαφή, θα πρέπει να είμαστε εντελώς αρνητικοί, ε, διότι ε, λειτουργεί σορευτικά όλη ε, όλος ο επηρεασμό στην ανθρώπινη υγεία από την συνεχή έκθεση σε αυτές τις ακτίνες και δεν γνωρίζω πόσοι από εμά αντιλήφθηκαν ότι την περασμένη Παρασκευή η Αρχή για την Ασφάλεια Μεταφορών των ΗΠΑ, η TSA, προχωρά σε μια εκτεταμένη ε, επανεξέταση των ε, σαρωτών σώματος, το σύνολο αυτών που έχουν εγκατασταθεί στα αμερικανικά αεροδρόμια, γιατί υπάρχει ε, εγνωσμένη αμέλεια στο σύστημα καταγραφής του επίπεδου ακτινοβολίας. νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε αν η αμφιλεγόμενη σχετική ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων δικαιολογεί βιασύνη ε, σε ένα θέμα που έχει τόσο κρίσιμες υπολογίες στη δημόσια υγεία. Και αναφέρομαι στην αποτελεσματικότητα, διότι η εμπειρία που είχαμε στην επίσκεψή μας στο αεροδρόμιο του Σίπχολ έδειξε ότι υπάρχει μια λυπής αποτελεσματικότητα. Θυμάμαι το κινητό στο παπούτσι του Μικέλε που πέρασε χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον Σαρωτή, ενώ αντιθέτως ο ένας από τους δύο που δοκίμαζαν το πέρασμά τους από, από το σαρωτή έπρεπε να ελεγχθεί, αφού έδινε false alarm, έπρεπε να ελεγχθεί στη συνέχεια με την κλασική μέθοδο της ψηλάφισης. Έτσι λοιπόν θέλουμε και διπλάσιο χρόνο και επιπλοκία στην ροή της, ε, ε, του όλου ζητήματος και τέλος υπάρχει και το αναπάντητο ερώτημα ποιος θα πληρώσει όλη αυτή την υπόθεση ε, που φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα πέσει και αυτό ε, στο κεφάλι των ε, επιβατών. Νομίζω ότι είναι ε, πολύ νωρίς. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα αναπάντητα για να υιοθετήσει και να προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την υιοθέτηση της γενικής εφαρμογής των σαρωτών σώματος. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ τον εισηγητή για την δουλειά που έχει κάνει. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται εδώ και χρόνια και περνάει από επιτροπή σε επιτροπή. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έχω ήδη πει. Ε, απλώς να τονίσω ότι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου όλοι είναι ότι αν δεν προσέχουμε και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουμε το κείμενο το οποίο θα υποβάλουμε. Λοιπόν, αν δεν είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, δεν θα ε, έχουμε την, ε, τους αρωτές σαν ε, το βασικό σύστημα ελέγχου ασφαλείας. Όταν πηγαίνεις σε ένα αεροπλά, αεροδρόμιο πρέπει να ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία ασφάλειας και να μην αρχίζει εκεί και αυτό θα πρέπει να είναι βασικό στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τους σαρωτές. Επίσης για το θέμα του κατά πόσον θα πρέπει να καταστρέφουμε αμέσως τις εικόνες. Ε, από τη στιγμή που τις παίρνουμε τις εικόνες και τις επεξεργαζόμαστε, οι εικόνες πρέπει να καταστρέφονται, δεν μπορούν να αποθηκεύονται. Έχουμε δει διάφορα ε, στο στοιχεία, στο χήθρο, διάφορες περι διάφορα περιστατικά όπου γίνεται κατάχρηση και κακή χρήση αυτών των ε, μηχανημάτων. Αυτό θα πρέπει να τιμωρείται. Κάτι άλλο ε, συμφωνώ με τον κύριο Βαντάλεν και με άλλους για το θέμα των ε, backscatter και της ε, τεχνολογίας ακτινογραφίας, ακτινοβολίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει δεκτό στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το λέω αυτό γιατί σήμερα μου ήρθε μια επιστολή που έχουν υπογραφή, ε, που έχει την υπογραφή τεσσάρων επιστημόνων από την ε, Εταιρεία Επιστημόνων στις Ηνωμένε Πολιτείε και ε, το υποσυπογράφηκε ο τεχνικός σύμβουλος του Προέδρου Ομπάμα. Αυτοί οι, επιστήμονες έχουν κάνει τέστα σε αυτή την τεχνολογία και λένε ότι οι δερματολόγοι και ε, ογκολόγοι, ειδικοί για τον καρκίνο, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες. Καταρχάς, ένας μεγάλος πληθυσμός ε, των, ε, των επιβατών πάνω από 65 χρόνια κινδυνεύουν από την ακτινοβολία γιατί μπορεί να δημιουργηθούν μελανόματα. Ε, επίσης, τα άτομα τα οποία είναι, ανασ... που ε, ε, είναι ανασοανοσιοκατασταλμένα. Ε, μπορούν να ε, υποστούν βλάβες από τα μηχανήματα αυτά. Επίσης, ε, κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρόκειται να διαβάσει όλη την επιστολή, αλλά τέλος πάντων αν ενδιαφέρεστε ρωτήστε τον βοηθό μου. Λένε στο τέλος αυτοί οι επιστήμονες ότι οι σαρωτές θα αυξήσουν τον κίνδυνο καρκινογέννηση στα παιδιά και άλλα μέλη ευαίσθητα και, και όλες οι ζημιές αυτές θα είναι δυσανάλογες με το όφελος που θα έχουμε για την πρόληψη των τρομοκρατικών ενεργειών. Επομένως, νομίζω ότι όλα τα επιχειρήματα για, την, για να μην χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία αυτή στην Ευρώπη βρίσκονται σε αυτή την επιστολή και ελπίζω ότι τα μέλη και η Επιτροπή θα λάβουν υπόψη του αυτού του είδους, υπόψη του αυτού του είδους αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί όταν υποβάλλουμε ε, τροπολογίες σε αυτή την ε, έκθεση και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω εάν ο κύριος ε, Πασκουάλ Ντεγκάντες έχει αυτή την επιστολή, έχετε διαβάσει την επιστολή αυτή. Όχι, όχι. Φίλιπ, μήπως μπορείς Α, μόλις ούτως ή άλλως σήμερα μόλις την πήρα και εγώ. Λοιπόν, μήπως μπορείς α, ε, να δώσεις και ένα αντίγραφο στον α, ε, εισηγητή. Ο κύριος Μπόλτουιν ε, εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω, είναι η πρώτη μου μέρα εδώ και είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να μιλήσω στην Επιτροπή σα και προσβλέπουμε ιδιαίτερη ευχαρίστηση στη μελλοντική μα συνεργασία. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Καταρχά να ευχαριστήσω τον κύριο Τεγκράντε Πασκουάλ για την πολύ ολοκληρωμένη και ισορροπημένη έκθεση. Ε, μας δίνει μια σαφή εικόνα σε εμά στην Κομισιό για το, για το πού βρίσκεται το Κοινοβούλιο και ποιες είναι οι απόψεις του για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και ελπίζω ότι θα έχουμε σοβαρέ συζητήσει και στο μέλλον για αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά του σαρωτέ, ε, εμείς πιστεύουμε ότι η απειλή είναι ε, πραγματική και το, μας το υπενθυμίσανε αυτό και τον Οκτώβρη όταν, κάποιος, όταν κάποιοι αποφάσισαν να ε, επιτεθούν στην πολιτική αεροπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει κίνδυνος. Και μετά το ψήφισμα του 2008 αναλύουμε γενικότερα την όλη κατάσταση. Είδατε την ανακοίνωση που κάναμε το 2010 και το καταλήξαμε σε κάποιες, σε κάποιες σαφείς απόψεις. Καταρχάς ότι οι σαρωτές είναι μια βάσιμη εναλλακτική λύση στα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζουμε τώρα, διότι ελέγχουν τα μεταλλικά και τα μη μεταλλικά στοιχεία και συμφωνώ βέβαια με πολλούς από αυτούς που πήρα το λόγο σήμερα ότι δηλαδή θα πρέπει να σέβονται συγκεκριμένα, συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα κριτήρια τα μηχανήματα αυτά. Καταρχάς, ε, είναι μηχανήματα που, τα, που γίνονται δεκτά από τους επιβάτες. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι θεμελιώδεις ελευθερίες, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ούτως ή άλλως όσον αφορά τους, τους, ε, τα μέτρα ασφάλειας ε, και τους ερωτές ε, στην, στα αεροδρόμια, η νομοθεσία είναι λίγο κατα, κατακαιρματισμένη. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια την προστασία των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων. Τώρα όσον αφορά την μελέτη σκοπιμότητας και των, και συνεπειών, η μελέτη αυτή θα ολοκληρωθεί και θα δημοσιευθεί πιο γρήγορα. Και υπό το φως της ανάλυσης που θα κάνουμε και υπό το φως των συζητήσεων που θα έχουμε και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα ε, προτείνουμε, θα υποβάλουμε προτάσεις μας για μια μελλοντική νομοθεσία τους επόμενους μήνες. Όμως θα πρέπει η νομοθεσία αυτή προφανώς να ε, συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένε ε, διατάξεις προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε για το φορτίο, για τα εμπορεύματα, για την ασφάλεια των εμπορευμάτων ε, ε, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Ξέρετε ότι έχουμε ε, σαφείς οδηγίες, αυστηρές οδηγίες ελέγχου για τον έλεγχο αυτών των εμπορευμάτων όσον αφορά αυτά τα οποία φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι αυτά τα οποία έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ο έλεγχος πρέπει να γίνει στην χώρα αποστολής. Εδώ υπάρχουν κάποιες αδυναμίες και ελπίζω ε, να θεωρήσετε ότι μετά τα περιστατικά του Οκτωβρίου απαντήσαμε γρήγορα διότι ε, έχουμε κάνει πιο αυστηρή, αυστηρό τον έλεγχο και ε, προσπαθούμε οι συστάσεις αυτές οι οποίες εκδόθηκαν να εφαρμοστούν κιόλας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Ντεγκράντες. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους έλαβαν το λόγο και πήρα μέρος στη συζήτηση. Να ευχαριστήσω και αυτούς που συμφωνούν με τις απόψεις μου και αυτούς που διαφωνούν. Γιατί σημειώνω ακόμη και τις διαφωνίες. Πάντως γενικά πιστεύω ότι από όλες τις παρατηρήσεις που ακούσαμε οι περισσότερες ή περιλαμβάνονται στη, στην έκθεση ήδη, είτε μπορούν να υποβληθούν και άρα να υποστούν κάποια τροποποίηση, βελτίωση μέσω των τροπολογιών που θα καταθέσετε και περιμένω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μόλις πριν από λίγο ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται την πρόταση, την παρότρινσή μας να θεσπίσει μια νομοθετική πρόταση για το θέμα αυτό. Βέβαια, βρισκόμαστε ακόμη στην αφετηρία μιας ε, προσπάθειας και ενός δρόμου που θα είναι μακρύς. Γιατί στα πλαίσια της συναπόφασης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Πριν από λίγο σας μίλησα για το ιστορικό και μάλιστα η ανακοίνωση που είχε δημοσιεύσει τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε χαρακτηριστεί από όλους μας ως ατελής και λυπής, γι' αυτό και την απορρίψαμε. Γιατί η ανακοίνωση αυτή δεν έλαβανε ε, τα απαραίτητα μέτρα για, την, ε, για το σεβασμό και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε τις επικρίσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπέβαλε μια νέα ανακοίνωση στην οποία καλύπτει τις προηγούμενες της αδυναμίες και μάλιστα συμπληρώνει επαρκώς ε, την προηγούμενη πρόταση, διασκεδάζοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες μας. Βέβαια, όπως λέμε σε όλες τις γλώσσες, το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Και είπα και μόνος μου ότι η κατάσταση σήμερα δεν είναι τέλεια και η πρόταση αυτή δεν είναι τέλεια. Θα ήταν όμως απαράδεκτο τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να αποποιηθούν των ευθυνών τους γιατί φέρουν την ευθύνη να συμμετέχουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντέδρασε, ανταποκρίθηκε στην ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπέβαλε παρατηρήσεις, συστάσεις που προσπάθησα εγώ να συμπηλήσω στην ε, έκθεσή μου. Προσπάθησα να καλύψω ένα σημαντικό φάσμα ε, σκέψεων και προτάσεων που μπορούν μεταξύ τους να συνδυαστούν. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι χρειάζονται μέτρα για αυτά. Και επίσης πιστεύω ότι επειδή υποχρεούμαστε να αναλάβουμε μια δράση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επειδή έχουμε τους αρωτές νέας γενιάς και εφόσον αυτοί τηρούν τη, τα θεμελιώδη δικαιώματα, δεν ε, καταστρατηγούν το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα και στην ιδιωτική ζωή. Από τη στιγμή που θα καταστρέφονται αυτόματα τα δεδομένα μέσως μετά την ε, χρήση της εικόνας, μετά τη λήψη της εικόνας. Και σίγουρα ε, το κείμενο θα πρέπει να υποστεί κάποιες διορθώσεις. Η αγγλική μετάφραση που διάβασα είναι προβληματική σε σχέση με το ισπανικό πρωτότυπο. Θα προτείνουμε την αυτόματη καταστροφή αυτών των εικόνων. Από τη στιγμή που ο επιβάτης θα περνάει από το σαρωτή, μετά θα καταστρέφεται αυτή η εικόνα που ελήφθη. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχει επιβλαβής επίπτωση στην δημόσια υγεία, στην υγεία των πολιτών. Αλλά από τη στιγμή που αποσοβήσουμε όλους αυτούς τους κινδύνους, είμαστε υποχρεωμένοι να δράσουμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Γιατί η έκθεση αυτή, όχι μόνο για τους αρωτές σώματος, έχει μετατραπεί σε ένα ευρύτερο θέμα, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία. Δεν μιλούμε μόνο για τους αρωτές σώματος, μιλούμε για τα υγρά, τα σπρέ λοιπά. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχει τεχνολογία διαθέσιμη, ας προχωρήσουμε. Και θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη. Εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς και να εμβαθύνουμε στην ανάλυση του θέματος. Είναι ένα θέμα πολύ λεπτό, όπως μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η τρομοκρατία χρησιμοποιεί μερικές φορές το ταχυδρομείο και τα φορτίο, την μεταφορά ε, εμπορευμάτων μέσω αεροπορικών μεταφορών για να υλοποιήσει κάποιες ε, τρομοκρατικές ενέργειες. Φυσικά δεν μπορούμε να αποσοβήσουμε οποιοδήποτε κίνδυνο, αλλά Εμεί εκπροσωπούμε του ευρωπαίου πολίτε. Οφείλουμε να μεταφέρουμε την ανησυχία του και να υποβάλουμε κάποιε προτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλε οι προτάσει που έγιναν νομίζω ότι έχουν τη θέση του. οι επικοδομητικέ τουλάχιστον, έχουν τη θέση του στην έκθεση αυτή. Βέβαια μερικοί είναι κάθετα αντίθετοι. Αλλά δεν μπορούμε απλώ να χρησιμοποιούμε ω άλοθη μερικέ θέσει ή να μιλούμε για τι αρνητικές συνέπειε των ακτίνων Χ, αφού ούτως ή άλλως το λέμε στην έκθεση, ότι αποφεύγουμε αυτή τη χρήση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί το συμβατικό σύστημα και την επιτροπολογία. Εμεί δεν διαλέγουμε το σύστημα. Θα ήταν υπερβολικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εγώ προτιμώ τα millimeter wave και εγώ προτιμώ ή την άλλη τεχνολογία, τους, α, τις ακτινοβολίες Θα ήταν εσφαλμένο κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τις ακτίνες χ, το σύστημα των ακτίνων που είναι συμβατικός τρόπο, και μάλιστα με τι ελάχιστε προδιαγραφέ και τι ελάχιστε τιμέ που προβλέπονται, σε περίπτωση που πουνε τα κράτη-μέλη, είπαμε ότι απορρίπτουμε αυτό το σύστημα, γιατί μερικοί αυτό λένε. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο σε σχέση με ορισμένε παρατηρήσει που ακούσαμε. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να αντιταχθούμε στο δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόσουν πιο περιοριστικά μέτρα. Όπως ισχύει και σήμερα. Γι' αυτό και έκανα και αυτή την επιφύλαξη. Ας έχουμε κάποιες ελάχιστες διατάξεις, αλλά ποιος μπορεί να αφαιρέσει από το Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα να υιοθετήσει αυστηρότερους κανόνες. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί πολύ πιο δραστικέ μεθόδου. Αλλά έχει δικαίωμα. Δεν μπορεί να αφαιρέσει κανένα στο Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ακτίνε χ, α πούμε. Λέω, α υιοθετήσουμε κάποιου ελάχιστου κανόνε. Και αν υιοθετήσουμε κάποια συμβατικά συστήματα θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Αλλά προσοχή, τα κράτη-μέλη δίνανται και έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν πιο αυστηρές διατάξεις, πιο περιοριστικά μέτρα. Κύριε Βαντάλεν, όσο αφορά τους ελέγχους, ανέφερα και τους ελέγχους στην έκθεσή μου, γιατί οι εμπειρογνώμονες που έχουν τεχνικές γνώσεις και γνωρίζουν το θέμα του φορτίου και των εμπερβατών είπαν ότι δεν γίνονται σοβαροί έλεγχοι στα φορτία που μεταφέρονται αεροπορικά. Και στο θέμα του φορτίου έχουμε πολύ περισσότερο δρόμο να διανύσουμε. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του φορτίου είναι έλεγχος ή επιθεώρηση. Θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Φυσικά με απόλυτο σεβασμό τη αρχή τη επικουρικότητα. Δεν πρόκειται εδώ να, να μπούμε σε χωράφια όταν δεν έχουμε αρμοδιότητα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλάβει κάποιε ευθύνε και αρμοδιότητε, θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην εξασφάλιση της πολιτικής αεροπορίας, αλλά με τα όρια των αρμοδιοτήτων της και με σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Εμείς ό,τι και να πούμε υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ισχύουν και οριοθέτηση αρμοδιοτήτων. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ ονομαστικά στους ε, ομιλητές και στα σχόλιά τους. Εγώ τα σημείωσα όλα καταλεπτός και νομίζω ότι από τη στιγμή που θα διατυπωθούν και τροπολογίες θα είναι δυνατό να καταλήξουμε και στις συμβαστικές λύσεις. Ακόμη και εγώ θα διορθώσω κάποια κομμάτια της εκθεσής μου, θα τα συμπληρώσω εφόσον υπάρχουν ανησυχίες από τους ευρωβουλευτές. Νομίζω, εφόσον εντάσσονται στον κανονικό μας στόχο, μπορούν κάλλιστα να βρουν τη θέση ε, στην έκθεση. Αλλά η θέση μου είναι σαφής, της α, ε, ανέλησα με εντυμότητα και σας είπα ποια είναι η γνώμη μου. Τώρα, οι σαρωτέ είναι ένα θέμα, τα υγρά είναι ένα άλλο θέμα, το φορτίο είναι ένα τρίτο θέμα. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τη ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία προσπάθησα να κάνω και μια πιο διεξοδική ανάλυση. Θα ήθελα να πω όμως ότι στα θέματα της καταπολέμησης τρομοκρατίας δεν μπορούμε να υπησερχόμαστε σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί υπάρχει και θέμα ε, εμπιστευτικότητας και απόρριτων πληροφοριών. Θέλουμε βέβαια την διαφάνεια, αλλά στην πολιτική δεν αναλύουμε τις στρατηγικές και συγκεκριμένες αποφάσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, εμπίπτουν και στην αρχή της εμπιστευτικότητας. Κάποιες αποφάσεις θα τις λάβουμε στα πλαίσια της επιτροπολογίας. Εμείς όμως θα χαράξουμε μόνο τις αδρές γραμμές που θα τις χρησιμοποιήσει ως πηγή έμπνευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να καταθέσει μια νομοθετική πρόταση και μετά να επανέλθουμε στη συγκεκριμενοποίηση αυτών των κανόνων και των διατάξεων και να φέρουμε σε αίσιο πέρας την προσπάθειά μας και να ανταπεξέλθουμε στις ευθύνε και τι υποχρεώσει μας. Σας ευχαριστώ κύριε Δεγκράντες. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών λήγει στις 21 Μαρτίου. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στη συνεδρίαση μας του Απριλίου. Τότε θα ψηφίσουμε στη συνεδρίαση του Μαΐου και στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. 21 Μαρτίου λοιπόν διορία για τις τροπολογίες, εξέταση των τροπολογιών τον Απρίλιο, ψηφοφορία στην Επιτροπή τον Μάιο και ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Σας ευχαριστώ. Πεντάλεπτη διακοπή για να εκενωθεί η αίθουσα και να περάσουμε στην κεκλεισμένα το θηρό συνεδρίαση των συντονιστών.